I think that we can uh, start. Ο πρόεδρος, ας αρχίσουμε λέει. Και. Α, να σας το πω στα Ιταλικά. Διότι για μένα είναι πιο εύκολο. Ε, βέβαια έχουμε κάτι να ε, κάνουμε κάποιε ερωτήσει στην Επιτροπή και θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι δεν θα εχουμε παρεξηγήσεις. παρεξηγήσει. Πρώτα-πρώτα, γι' αυτό σας λέω θα πρέπει να δω τι γίνεται με την Κομισιόν και κατά πόσον ε, υπάρχει συμφωνία ούτως ώστε να προσθεθεί αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη για τη σημερινή ε, συνεδρίαση. Είναι κάτι το οποίο προσθέθηκε ετήσι πολλών πολιτικών ομάδων και ε, έχει να κάνει με αυτά τα τελευταία σκάνδαλα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εγκρίνει τη καινούργια διαδικασία Real Driving Emissions και αυτό σε τέσσερα πακέτα. Πρώτα-πρώτα ε, αυτά τα πρώτα μέτρα εγκρίθηκαν στις 19 Μαΐου και επίση είπαμε ότι έτσι ξεκίνησε η σύνταξη αυτού του μέτρου και αυτό μέσω της ε, επιτροπολογίας. Κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται ε, σύντομα να αναδειχθεί αυτό το νομοθέτημα αλλά δεν είχε εμπλακεί το Κοινοβούλιο. Οπότε και εμείς αυτό το οποίο τώρα θέλουμε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει πώς έχουν τα πράγματα και πώς προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ούτω ώστε να αποφύγουμε ότι αυτές οι απλές διαδικαστικές μεταβολές είναι δυνατόν να μας οδηγήσουν σε μια δεύτερη τέτοια φάση κατά την οποία πάλι να μην εμπλέκεται το Κοινοβούλιο στη διαδικασία και για αυτό το λόγο απευθυνόμαστε στην Επιτροπή και θέλουμε να τη ζητήσουμε να μας ενημερώσει πριν εγκριθούν αυτά όλα τα μέτρα με την Επιτροπολογία, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει αυτή την δυνατότητα να υποβάλει τις ε, τυχόν ενστάσεις του όσον αφορά τα όσα συζητούνται τώρα. Οπότε και ευθύ αμέσω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκουέν Κοζιγκό, τον πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή για να μας εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την ε, διαδρομή, τη διαδικασία αυτή που θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και κατόπιν βεβαίως πρόκειται να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για αν θέλουν ούτως ώστε να υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, σύμφωνα με τις διατάξεις ε, του σχετικού κανονισμού για τα όρια των εκπομπών από τις εξαρμίσεις ε, συμφωνήθηκαν οι φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και έχουμε κάποιες διατάξεις που ε, ορίζονται από το EDC βάσει συγκεκριμένων δοκιμών από το 2011 ασχολούμεθα για να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες δοκιμών ούτως ώστε αυτά τα περίπλοκα τεστ να συμπληρωθούν και έτσι να μπορούμε να κάνουμε τη μέτρηση των πραγματικών εκπομπών κατά την οδήγηση. Πρώτο βήμα έγινε τον Μάιο με αυτόν τον κανονισμό ο οποίος ε, τώρα ε, επανεξετάζεται για να δούμε ποιο θα είναι το εφαρμοστείο σύστημα αυτό το σύστημα το οποίο συζητούμε και τώρα βρισκόμαστε ήδη στην προετοιμασία της δεύτερης φάσης ούτω ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε το ποιες θα είναι οι οριακές τιμές οι οποίες θα ισχύσουν σύμφωνα με ε, αυτές τις νέες δοκιμές και έτσι η κατάσταση να προσαρμοστεί στον αρχικό κανονισμό και έτσι να έχουμε τις φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για ε, αυτού του είδους τις μετρήσεις και να μην έχουμε κάποια άλλες τεχνητές ε, τιμές και οπότε είχαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν άσχετα με αυτό το οποίο γινόταν στον δρόμο. Και όπως τα γνωρίζετε, οι συνομοθέτες που αποφάσισαν αυτή η προσαρμογή των ε, δοκιμών να καταλήξει σε κάποιο είδους καθορισμό οριακών τιμών. Μόλις οριστούν οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες ε, της μέτρησης και αυτό να γίνει με επιτροπολογία και αυτό και κάνουμε τώρα. Ούτως ώστε να θεωρήσουμε ότι 6 Οκτωβρίου ήρθαμε σε επαφή με το Συμβούλιο για το τι προσέγγιση θα γίνει, τι προβασκευαστικό έργο θα γίνει και επίσης πριν τα τέλη του μηνός αυτού πρόκειται να ξανασυνδυθούμε και γι' αυτό και λέμε για τις 28 δεκάτους. Επίσης Θέλουμε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Βεβαίω και θα κινηθούμε στα πλαίσια της διοργανικής συμφωνίας. Προβλέπεται κάποια διάρθρωση της ε, διαδικασίας και αυτό και απεφάσισαν οι συνομοθέτες όταν ε, ε, ενέκριναν το σχετικό κανονισμό και μετά την πρώτη αυτή συζήτηση, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια πρώτη αντίδραση από τα κράτη-μέλη για το τι πρεσβεύουν. Οπότε και τους είπαμε στις 16 Δεκάτου να μας αναφέρουν σχετικά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ετοιμάσει τη σχετική πρόταση η οποία θα σας διαβιβαστεί και ταυτόχρονα θα αποσταλεί και στα κράτη-μέλη. Μόλις επομένως έχουμε αποκρισταλώσει τη θέση μας. Τώρα, ο συνάδελφο μπορεί να συνεχίσει. Δύο-τρία λόγια κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σα πω γιατί την ακολουθητή διαδικασία. Διότι όπω θα ενθυμίστε, είχαμε την εισαγωγή αυτών των ε, δοκιμών, αυτών των τεστ για τις real driving emissions, τις πραγματικές, ε, ε, τα, τα πραγματικά καυσέρια τέλο πάντων, με πραγματικές συνθήκες. Και αυτό κατέκρισε έναν κανονισμό ο οποίο εγκρίθηκε από μια επιτροπή εκπροσώπων των κρατών μελών τον Μάιο και ευθύς μετά την έγκριση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε το κείμενο αυτό το οποίο προήλθε από το έργο της Επιτροπής εκείνης. Είχαμε επίσης ε, το σύνολο των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών και επίσης και τα πρακτικά των συζητήσεων. Οπότε ε, αυτό το πρώτο νομοθέτημα υπόκειται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα δε με τον κανονισμό για την επιτροπολογία, το Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει αυτές τις νομοθετικές πράξεις και να δει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε στα πλαίσια της εντολής της για τις ε, ε, εφαρμοστικές της ε, αρμοδιότητες. Όπως είπε ο συνάδελφος, θα καταλήξουμε σε κάποιο είδους οριακές τιμές, θα υπάρξει κάποιο χρονοδιάγραμμα και ο στόχος μας είναι να γίνει η ψήφιση στην Επιτροπή στις 28 Δεκάτου. Όμως το κείμενο της ε, προτάσεως πρόκειται να ανέβει στο σχετικό site για την Επιτροπολογία ακριβώς μόλις θα είναι έτοιμο την Επιτροπή και θα διαβαστεί ταυτόχρονα σε κράτη-μέλη και εις Κοινοβούλιο. Και μόλις ψηφίσει η Επιτροπή, ελπίζουμε αυτό να γίνει στις 28 Οκτωβρίου, πρόκειται να λάβετε μια σύνοψη της συζητήσεως και επίσης τα συνολικά αποτελέσματα της ε, ψηφίσεως. Στη συνέχεια δε πρόκειται να υποστεί το κείμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο όσον αφορά το εάν ετήρησε η Επιτροπή τις εφαρμοστικές της αρμοδιότητες. δει το λόγο άλλος κύριος από την Επιτροπή για να συμπληρώσω. Για να συμπληρώσω τα στοιχεία αυτά η συζήτηση για τους παράγοντες ε, συμμόρφωσης θα γίνει με τα κράτη-μέλη προτού οριστικοποιηθούν οι κανόνες για τα θέματα αυτά. Η Κομισιόν φυσικά ήθελε να εισαγάγει τα αποτελέσματα αυτά στη νέα, νέα διαδικασία το ταχύτερο δυνατό χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πραγματικές απαιτήσεις. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τεχνικής εφικτότητος και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένας σαφής δρόμος για πλήρη συμμόρφωση κάτω από, φυσιολογικά κάτω από σωστές και πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτό θέλουμε, δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα την πρότασή μας και όταν είναι έτοιμη θα επανέλθουμε σε εσά και τα κρατη Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Και θα δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Γκρότε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συζήτηση και έχουμε την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Γιατί πρέπει σε τελική ανάλυση να συμφωνήσουμε αν θα δεχτούμε διαδικασίες επιτροπολογίες ή όχι. 28 Οκτωβρίου θα πρέπει να καταλήξουμε λοιπόν σε μια τελική απόφαση και νομίζω ότι και η δική μου ομάδα και πολλοί άλλοι κοινοβουλευτικοί θέλουν να ξέρουν το εξή. Αυτά τα οποία γίνονται τώρα στην δοκιμασία των αυτοκίνητων δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα οποία εκπέμπουν στους δρόμους. Ούτε η κατανάλωση, ούτε η εκπομπή ρήπων, σωματιδίων, οξυδίων του αζότου και τα λοιπά. Πώς θα γίνει λοιπόν το τεστ στο μέλλον για να είναι σε πραγματικές συνθήκες. Και σας υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια είχε θέσει το θέμα αυτό ο κ. και υποβάλει κάποιες προτάσεις για τις οποίες αξίζει να συζητήσουμε πώς θα εφαρμόσετε αυτό τον κανόνα των ε, ε, συνθήκων συμμόρφωσης. Υπάρχει ο παράγων αυτός ο οποίος ισχύει με κιλοβατο, κιλοβατόρες στα φορτηγά. Τι θα γίνει με τα μικρά αυτοκίνητα όμως, με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πώς μπορούμε να έχουμε μια χοντρική τέλος πάντων ε, ιδέα για το πώς θα καταλήγεται στα τελικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας και τους παράγοντες της συμμόρφωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ηγέρθηκαν με το σκάνδαλο των εκπομπών. Δεν έχουμε τεχνικές γνώσεις, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά, αλλά σε εσά να απόχετε να εξασφαλίσετε ότι η συμπεριφορά του αυτοκίνητου στον δρόμο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και τις εκπομπές ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία βρισκόνται στα διαφημιστικά φυλάδια των αυτοκινητοβιομηχανιών. Βλέπουμε να υπάρχει λοιπόν μια τεράστια σύγκρουση σε ό,τι αφορά τους στόχους. Από τη μία μεριά θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε την προστασία του κλίματος. Αυτό θα γινόταν ίσως αν είχαμε 100% ανανεώσιμες ενέργειες και 100% ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα των σωματιδίων που εκπέμπονται. Οι πραγματικές λοιπόν τιμές του τι εκπέμπει ένα αυτοκίνητο, το τι αναπνέουμε από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, είτε είμαστε στη Ρώμη, είτε είμαστε στις Βρυξέλλες, στο Χόλμη ή οπουδήποτε άλλο, είναι φανερό ότι αυτά είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία επιτρέπονται. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχει λάβει κανείς υπόψη αυτό. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το κλίμα και γι' αυτό πάρα πολλοί κατασκευαστές εστράφησαν προς το δίζελ. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τους στόχους μας σε ό,τι αφορά τη ρήπανση γιατί εκπέμπονται περισσότερα σωματίδια και περισσότερα οξύδια του αζότου. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς εσείς θα δημιουργήσετε αυτό το παράγοντα ε, ε, το λεγόμενο παράγοντα ε, συμμόρφωσης των αυτοκινήτων κατά πόσο θα λάβετε υπόψη τις ακραίες συνθήκες και κατά πόσο όχι, ώστε να μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των τιμών που καταμετρώνται στις δοκιμές και των τιμών που ισχύουν στον δρόμο. Και κατά τα άλλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και για το γεγονός που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Herr Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μ' αρέσουν τα πειράματα. Μ' αρέσει να είμαι σε επαφή με την εκλογική μου περιφέρεια. Οπότε εποφελήθηκα αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είχε γενέθλια και πάρτι ο 9χρονος γιος μου. Είχα λοιπόν μελλοντικού ψηφοφόρους που σήμερα είναι 9-10 ετών. Τους ρώτησα λοιπόν, αν θέλουμε να γνωρίζουμε τις πραγματικές εκπομπές ενός αυτοκινήτου, τι θα έπρεπε να οργανώσουμε. Μετά από πέντε λεφτά ήρθαν με ένα κοινό σχέδιο και είπαν αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να οδηγήσετε στο δρόμο ένα αυτοκίνητο και να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό εξοπλισμό μέτρησης των εκπομπών, οπότε θα ξέρετε ποιες είναι οι πραγματικές εκπομπές αυτού του οχήματος. Και πραγματικά ήταν μια εκπληκτική λύση ε, επιστημονική πραγματικά από νέα παιδιά. Και έτσι έμαθα τον Ιανουάριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε με μία σε βάθος ανάλυση ακριβώς επί αυτού του θέματος. Πώς δηλαδή να μετρήσουμε τις πραγματικές εκπομπές ενός οχήματος. Και μετά από λίγο λοιπόν καταλήξαμε στο ότι το όχημα θα ε, μετριότανε βάση φορητών, ε, δηλαδή ακριβώς αυτό που είπα τα 9 χρόνια και τα 10 χρόνια σε 5 λεφτά, οι άλλοι έκαναν 4 χρόνια να μας το πούνε. Αλλά εντάξει, το Μάιο του 2015 οι χώρες μέλη συμφώνησαν επιτέλους. Και μετά μας πήρε άλλους 7 μήνες να εφαρμόσουμε αυτές τις δοκιμές, αυτές τις μετρήσεις. Και ίσως ακριβώς επειδή είναι τόσο προηγμένη επιστήμη, ε, χρειάζεται και άλλος χρόνος για να αποφασίσουμε αν είναι όντω σωστό για να το εφαρμόσουμε. Ίσως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε αν δεν πρόκειται για πίεση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες των χωρών μελών, τότε γιατί παίρνει τόσα χρόνια να καταλήξουμε σε μια τόσο απλή λύση. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, έχω την αίσθηση ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχουμε μία που είναι με διαφάνεια, δημοκρατική, με λογοδοσία, όπου συμμετέχει το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορίζουμε ανώτατες τιμές εκπομπών είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Παράλληλα όμως έχουμε και μια άλλη διαδικασία μη δημοκρατική και μυστική όπου φαίνεται ότι το βασικό είναι πώς θα παρακάμψουμε την άλλη τη δημοκρατική διαδικασία. Και αυτή η δεύτερη διαδικασία είναι της Τεχνικής Επιτροπής. Όπως συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την Επιτροπή ακριβώς αυτή την υπόθεση της Volkswagen, συγχρόνως συνεδρίαζε στις Βρυξέλλες η Τεχνική Επιτροπή. Και εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει ακόμα πρόταση. Αλλά από τις δικές μου τις πληροφορίες κάτι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει πρόταση με 1,6 δίκτυο 2017 και το 2018, δίκτυο συμμόρφωσης, και 1,19 μετά από το 2019. Όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα που δεν είναι δυνατό να πρόκειται για μη πρόταση. Είναι θέμα βέβαια διατύπωσης. Μπορείτε να το πείτε non-paper. Εδώ όμω πρόκειται για μια πραγματική πρόταση που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τεχνική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς λοιπόν έρχεται και λέτε ότι όταν θα γίνει η πρόταση τότε θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει πρόταση. Μην χρησιμοποιούμε τώρα λάθος διατυπώσεις και λέτε ότι δεν υπάρχει πρόταση. Υπάρχει πρόταση. Και ρωτάω. Εφόσον δεν υπάρχει διαφάνεια και από εκεί απορρέει το πρόβλημα με τη Volkswagen, μήπως θα έπρεπε να τροποποιήσετε την πολιτική σας όσον αφορά τη διαφάνεια. Σήμερα στους Financial Times κάποιοι επενδυτές, πάνω από 600 δις ε, Λύρε. Ακριβώ αυτό λένε. Λένε ότι θέλουν διαφάνεια γιατί φοβούνται ότι διακυδεύεται εδώ η ίδια εξοπιστία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξετε την πολιτική σα για τη διαφάνεια. Και εσεί λέτε ότι θέλετε πλήρη διαφάνεια, αλλά μετά έρχεται και συνοψίζετε την συνάντηση σε δύο γραμμέ. Εγώ θέλω πλήρη διαφάνεια. Θέλω την πρόταση λοιπόν να έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω επίσης όλες τις θέσεις των χωρών μελών. Θέλω να ξέρω τι λέει κάθε μία. Δεν νομίζετε ότι στην κρίση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για την ποιότητα του αέρα πρόκειται και πάνω 500 εκατομμύρια ανθρώπους δεν έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν οι εθνικές τους κυβερνήσεις, εκ μέρους τους, τι θέσεις υποστηρίζουν, αλλά να γίνεται αυτό πίσω από κλειστές πόρτες. Αν κάποιες χώρες θέλουν τρία ε, δείκτης παράγοντας η μόρφωση. Στο το κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας το πείτε. Τέλος, Πρόεδρε, για το κατά πόσο ναι ή όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγνώριζε τα προηγούμενα. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την Επίτροπο 200 και είπε ότι η Επιτροπή δεν τα γνώριζε. παρά τις εκθέσεις του 2011 και του 2013. Εγώ όμως δυσκολεύομαι να αντιληφθώ το εξή. Στις εκθέσεις αυτές δεν αναφέρονται ρητά αυτοί οι εξοπλισμοί εξαπάτησης, αλλά δεν νομίζετε ότι ακριβώς είναι ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν κυκλοφορούν ιδέες ότι υπάρχουν τέτοιοι εξοπλισμοί να ρωτήσει τις χώρες μέλη για το πώς εφαρμόζουν τους κανόνες και να εξηγήσουν γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δοκιμές που γίνονται στα εργαστήρια και τις άλλες. Εξηγήστε μου λοιπόν σας παρακαλώ πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν το έκανε, γιατί δεν απευθύνθηκε στις χώρες μέλη και όλα αυτά. Ευχαριστούμε κύριος Εκχαουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριο Χερπράντη. Νομίζω ότι η Κομισιόν συνεχίζει με το business as usual, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Σαν να ήταν οι πολίτες σε μια κατάσταση που δεν θέλουν να ξέρουν τι έγινε, που δεν τους νοιάζει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να μην θέλουν να ξέρουν τι κάνουν τα κράτη-μέλη του. Εξακολουθούν να έχουν αυτή τη μυστικοπαθή προσέγγιση λέγοντα «Μα δεν υπάρχει μια επίσημη πρόταση ακόμα». Μα για σταθούμε, για σταθείτε μια στιγμή. Πρέπει να είμαστε τίμοι προ του πολίτες μας. Έχει, υπάρχει μια εξαπάτηση. Αυτό το θέμα είναι υπό επεξεργασία εδώ και πολλά χρόνια και οι πολίτε μα αξίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια από την Κομισιόν. Τι προτείνει η Κομισιόν, τι θέλουν τα κράτη-μέλη. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρόταση Κομισιόν που έχει κατατεθεί. Αλλιώς γιατί ζητάτε από τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν πριν από την Παρασκευή. Σε τι αντιδρούν άμα δεν έχετε καμία πρόταση. Έχετε προτείνει αριθμούς όπως και το 1,6 ως παράγοντα συμμόρφωσης. Δηλαδή διαφορά μεταξύ σχέση μεταξύ πραγματικών και ε, τιμών που μετρώνται στο εργαστήριο. Μα η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθείτε εσείς ως Κομισιόν να είσαστε μυστικοπαθείς για τις προτάσεις της δικές σας. Δεν τολμάτε να πείτε στους πολίτες τι προτείνετε εσείς και τι κάνουν τα μελη Μιλάτε για μια διαθεσμική συμφωνία. Αλλά ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι το Κοινοβούλιο να παίρνει μαζί με τις επιτροπές του Συμβουλίου όλα τα μέτρα τα οποία προτείνονται για εφαρμοστικά θέματα και τις σημαίες διατάξεις των ειδικευμένων επιτροπών. Εμείς θέλουμε διαφάνεια για αυτά που προτείνετε και θέλουμε ότι πρέπει να μας δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο και αυτό σας δίνει πολύ περιθώριο να πείτε, να εξηγήσετε τι θέλει το Συμβούλιο. Μόνο έτσι μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αυτό το απαιτούμε όχι εμείς, αλλά οι πολίτες μας. Και δεν θέλω να ακούσω άλλα φορμαλιστικά επιχειρήματα όπως αυτό δεν είναι ακόμα επίσημη πρόταση. Κανείς δεν το καταλαβαίνει αυτό. Υπάρχει μια πρόταση, έχει σταλεί στα κράτη-μέλη. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να δώσουν μια απάντηση. Στείλτε το και στους υπόλοιπους για να καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά για τη διαφάνεια. Και τώρα για το 1,6 ως παράγοντα συμμόρφωσης. Το μόνο που μπορώ να συμπεράνω από αυτόν τον παράγοντα συμμόρφωσης είναι ότι το όριο των 80 μιλιγκράμμ το πολλαπλασιάζεται από 1,6. Μπορεί κανείς να εκπέμπει περισσότερα από 80 mg τα οποία περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Και θα ήθελα να έχω και νομική αρρωγή και από εσά και από εμά. Στο άρθρο 5.1 λέγεται σαφώς ότι θα πρέπει το αυτοκίνητο να συμμορφώνεται σε κανονικές συνθήκες με αυτόν τον κανονισμό και τις εφαρμοστικές του συνθήκες. Με αυτόν τον κανονισμό είναι σαφές, σημαίνει 80 mg. Τώρα έχετε μία εφαρμοστική διάταξη που το, το 80 γίνεται 128 mg. Αλλάζετε λοιπόν τους κανόνες του παιχνιδιού. Αντί για 80 μιλιγκράμμ πάτε στα 128. Με μία εφαρμοστική ρήτρα λοιπόν αλλάζετε ένα κομμάτι ενός κανονισμού. Μα είναι αυτό νομικά δυνατό. Εμείς έχουμε εγκρίνει ένα νομικό εργαλείο, ένα κανονισμό ο οποίος θέτει σαν όριο τα 80 μιλιγκράμμ τέρμα. Δεν καταλαβαίνω πώ εσεί με ένα εφαρμοστικό μέτρο μπορείτε να αλλάξετε την ουσία ενό κανονισμού. Και τέλο και αυτό είναι το τρίτο σημείο, θα πείτε ναι πρέπει να είναι τεχνικά εφικτό. Αυτή ήταν και η δική σα διατύπωση. Εδώ υπάρχουν κάποιε μελέτε που είναι ήδη από πέρσι που δείχνει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα στο δρόμο που ικανοποιούν αυτά τα πρότυπα. Τα ικανοποιούν. Είναι τεχνικά εφικτό να το κάνουν αυτό. Το ξέρουμε το ξέρουμε ότι οι διάφοροι κατασκευατές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες. Και ξέρουμε ότι οι ίδιοι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν άλλη τεχνολογία στην Αμερική και άλλη τεχνολογία στην Ευρώπη. Και αυτό γίνεται μονάχα για λόγους κόστους και κέρδους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεχνολογίες αυτές οι οποίες είναι ικανοποιητικές και οι οποίες μπορούν να σεβαστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακόμα και τα αμερικάνικα πρότυπα που είναι ακόμα πιο αυστηρά. Γιατί λοιπόν στο Λύκο συζητάμε εδώ τώρα για θέματα εφικτότητος. Μιλάτε για πιο ευέλικτους στόχους, κάτι το οποίο αντίκειται με τον, στον κανονισμό. Γιατί λέτε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό αυτό το πράγμα. Διαβάστε αυτές τις ε, έρευνες. Είναι τεχνικά εφικτό. Αν δεν θέλει αυτοκίνητο βιομηχανία, αυτό δεν είναι το θέμα. Μπορούν να το κάνουν όμως. Και δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά κόστους. Μπορούν να το κάνουν και είναι καιρός να είμαστε λιγάκι πιο σκληροί με αυτού που δεν θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν και είναι τεχνικά εφικτό. Και ίσω και η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί κάπως διαφορετικά εάν θέλει να έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη από την πλευρά των πολιτών. Thank you very much. And now... πάρα πολύ. Ο Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν τα ακούμε αυτά και βρίσκεται κανείς χρόνια εδώ στο κοινοβούλιο, αναρωτιέται, μα με τι ασχολούμαστε. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι εφικτό. Άκουσα και τους συναδέρφους, αλλά και εγώ έχω μιλήσει και με το γιο μου και με την κόρη μου. Είναι εύκολο να γίνουν αυτές οι δοκιμές, είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζονται συνεδριάσεις χρόνια και χρόνια, μπορεί να γίνει πολύ απλά. Στην Ολλανδία έχω καταλάβει από την πολιτική, από τον Υπουργό εκεί, ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα θέλουν να προχωρήσει η ρύθμιση. Οπότε εδώ γιατί να περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρόκειται για την υγεία μας. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί έχουμε ασχοληθεί και με τη γεωργία, με το μονοξίδιο του αζότου. Και εκεί έχουμε ζήτημα. Και εκεί αν εκεί γίνονται παραβιάσεις, τότε πρόκειται για πολύ σοβαρή απάτη κατά του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν βλέπω γιατί εδώ να μην μπορούμε να το κάνουμε. Όσο γίνεται πιο γρήγορα λοιπόν να εφαρμοστούν αυτά και να προχωρήσουμε. Και τέλος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κεντρικά κάποιο υπεύθυνο από την Ευρώπη που να πηγαίνει σε κάθε εθνικό κέντρο τέτοιων ελέγχων. Δεν θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο, θέλω όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσουμε με τη ρύθμιση και να προχωρήσουμε παρακάτω έτσι. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντάλη τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που ήρθε και μας ενημέρωσε. Αλλά, με όλο το σεβασμό, ισχνότατα είναι αυτά που μας είπανε. Μας είπατε δεν έχει οριστικοποιηθεί το τι θα κάνετε και είπατε ο αμιλητή θα ολοκληρώσετε το έργο σας, αλλά δεν μας είπατε το πότε. Και είδαμε τους ε, ε, συντελεστές να έχουν πρόταθεί. Μα γιατί δεν έρχεστε εδώ να μας τα πείτε με διαφάνεια και να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε το παράδειγμα παραθυμόν 1 στη σελίδα 9 όπου εκεί μας λέει το πώς γίνεται ο υπολογισμός. Όμως εμείς χρειαζόμαστε κάποιο είδους διαβεβαίωση. Με τι συντελεστή θα γίνουν όλα αυτά. Τι θα συμφωνηθεί. Μας λέτε ότι θα, θα κοιτάξετε την ελάχιστη οριακή τιμή, οπότε αυτό θέλουμε κι εμείς. Για πέστε μας ότι θα υπάρχει κάτι πάνω από το 1,5 σαν, παράνομα, σαν παράγον συγγνώμη, ε, ε, τήρησης του νόμου οπότε και, και κάπου να προκύπτει ότι χρειάζεται να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Κάτι άλλο τώρα. Σωστό το να μας διαβεβαιώσετε ότι αυτός ο συντηρητής συμμόρφωσης δεν θα είναι παραπάνω από αυτό το οποίο λέει ο κανονισμός δηλαδή 8 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Κάτι το οποίο θέλουμε να ε, σχετίζεται με την φυσιολογική οδήγηση. Γιατί μιλάμε τώρα για κανονισμό προ οκταετίας που τα είπε όλα αυτά, μα πολύ καιρό πέρασε. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, σήμερα μας είπατε για χρονοδιάγραμμα, όμως το Κοινοβούλιο ζητεί για φιλόδοξη και ταχεία διαδικασία εφαρμογής της, ε, της διαδικασίας των τεστ RDA. Όμως, πότε θα τηρηθεί αυτό που συμφωνήθηκε στην 1η Ιουλίου για το TCMV, οπότε είπαμε ότι ό,τι καθορίσει το σχονοδιάγραμμα θα πρέπει να εξεταστεί και να τηρηθεί. Είπαμε επίσης για κάποια εποπτική αρχή, εποπτική ρυθμιστική αρχή και είπαμε ότι θα γίνει μια πρώτη συνάντηση τώρα που ξέσπασε το σκάνδαλο Volkswagen. Σύμφωνοι, εσείς έχετε την αρμοδιότητα ε, πρότασης των κονισμών αρχή της εφαρμογής τους, γιατί έχουμε τις αρχές της εποπτείας των ε, εθνικών αγορών και τους ελέγχους στα αυτοκίνητα. Όμως οι εθνικές αρχές ούτε μπορούν ούτε ξέρουν να τα κάνουν όλα αυτά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια ευρωπαϊκή εποπτική ρυθμιστική αρχή μια αρχή που να μπορεί αυτά να τα χειριστεί. Thank you Now... Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ήβο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Όμως είναι σημαντικό και συμφωνώ με αυτά που είπαν η κυρία Νταλή και η κυρία Σχρέερ ότι μια ανεξάρτητη αρχή είναι αναγκαία ώστε οι δοκιμές να μπορούν να γίνονται με έναν ελάχιστο δίκτυ συμμόρφωσης. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία. Όχι θα λέγα εγώ. Διαθέτουμε μέσα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να είναι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι άλλο, αλλά πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή, υπερεθνική δηλαδή, που θα παρακολουθεί, που θα ελέγχει. Αλλιώς δεν έχουν νόημα όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Η Επίτροπος Διακόφσκα την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε στην Ολομέλεια δεν απέκλεισε, δεν το επιβεβαίωσε, αλλά δεν το απέκλεισε πάντως να γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τις δοκιμές RDE σε πραγματικές δοκιμές, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες αυτό που χρειάζεται είναι η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν. Οπότε θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει υπάρχει αυτή η δέσμευση επίσημα να υπάρξει μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή και να αποτελέσει αυτή μέρος του πακέτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στην Κομισιόν. Α, μια στιγμή. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντησα το λόγο, αλλά μόνο δεν με είδατε. Πάντως, ήθελα κάτι να σας πω. Γιατί, διότι ε, να μας πει η Επιτροπή από πού και σπου τώρα ενώ υπάρχουν ε, στοιχεία ε, και κατά την προηγούμενη ολομέλεια πάρα πολλοί συνάδελφοι λέγανε ότι έχουμε από το κοινό κέντρο ερευνών Υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις διάφορες ε, οριακές τιμές των καυσαρίων ότι υπάρχει software το οποίο έχει μπει στα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα στοιχεία και οι ενδείξεις επιβεβαιώθηκαν γιατί έγινε και παρουσίαση ολόκληρη από υπάλληλο της Κομισιόν ότι υπάρχουν τέτοιες συσκευές, τέτοιο software στα αμάξια και ότι επομένως ξεγελούσαν τα τεστ τα ευρήματά τους. Και αναρωτιέμαι, άπαξ και τα ήξερε αυτά η Κομισιόν ότι υπάρχει τέτοιο software από πού και που δεν ενήργησε γέρος και κυρίως τη στιγμή που προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, τι θα κάνουμε με εσωτερική αγορά και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδους θεμητές συνθήκες ε, ανταγωνισμό στην αγορά αυτή και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες όμως απίλαβαν ε, προτιμησιακής μεταχείρισης από τις αρχές. Οπότε, επομένως, δεν δόθηκε σημασία στην αγορά. Παρά τις δυσκολίες του να περιφρουρήσουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει μεταξύ εθνικών αρχών της τυποποίησης με τα εθνικά συμφέροντα των ε, αυτοκινητοβιομηχανιών. Τι θέλω να πω. Ότι πάρα πολλές από τις συγκρίσεις της Κομισιόν προέρχονται από το Λουξεμβούργο, από την αρχή του Λουξεμβούργου, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα σχετικό έγγραφο από κάποια μη κυβερνητική οργάνωση. Πολλές, πολλές τέτοιες άδειες από το Λουξεμβούργο. Μα τι γίνεται, αυτό επηρέασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να ξαναδώσουμε τον λόγο στην Κομισιόν. για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Παρακαλώ. Ίσως πρέπει να τα δούμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Μετά από τα πρόσφατα γεγονότα παρακολουθούμε διάφορες κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία, τα πραγματικά γεγονότα. Να υπάρξει συντονισμός των ερευνών όλων των ε, κρατών μελών που κάποια από αυτά κάνουν και διορθωτικές δράσεις. Έχουμε σε στόχο να έχουμε μια επαφή με τις αρχές των κρατών μελών μεθαύριο στις 15 του μηνός για να ξέρουμε τι έχει προκύψει από τις έρευνες που έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις έρευνες εμείς, αλλά μπορούμε σίγουρα να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριού μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των δράσεών μας. Και γίνονται φυσικά και διορθωτικές δράσεις. Το δεύτερο είναι αυτά που κάναμε για τις πραγματικές εκπομπές στο δρόμο. Το δεύτερο πακέτο και το τρίτο πακέτο θα είναι η εξέταση τα συστήματα έγκρισης κυκλοφορίας σε διάφορες αγορές έγκρισης τύπου δηλαδή. Αυτό λοιπόν για να ξέρετε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία της συνολικής μας προσέγγισης. Για το ερώτημα αν ξέραμε κάτι για όλα αυτά που έγιναν. Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν συσκευές οι οποίες μπορούν να παρακάμψουν και να εξαπατήσουν τη δοκιμασία. Ήδη από την νομοθεσία του 2007 ξέραμε ότι υπήρχαν και είχαν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν είχαμε όμως καθόλου πληροφορίες για την περίπτωση της Volkswagen στις ΗΠΑ από την Αμερικανική Υπηρεσία Αποστασίας του Περιβάλλοντος, την EPA. Ήρθαμε σε επαφή με την EPA μόλις μάθαμε από αυτούς ότι κάνουν αυτές τις έρευνες και σε σχέση με τις μελέτες των κοινών κέντρων ερευνών αντίθετα από ό,τι αναφέρεται, δεν ήταν κομμάτι των μελετών το να δουν αν υπάρχουν ή όχι τέτοιες συσκευε εξαπάτησης. Απλώς εξετάζαν αν οι, συσκευε αν συσκευές εξαπάτησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά οι μελέτες αυτές παρουσιάστηκαν στα κράτη-μέλη και όπως είπα προηγουμένως απαγορεύονται έτσι και αλλιώς αυτές οι συσκευές από τον κανονισμό μας. Βέβαια η εφαρμογή είναι θέμα των κρατών μέλων. Ήμασταν... Καθυστερήσαμε στην εφαρμογή τώρα ή όχι. Μετά από τις μελέτες αυτές που έγιναν το 2007 ξεκινήσαμε μία μελέτη για τα τεστ ε, οδήγηση στον δρόμο. Τώρα πείτε ότι είναι απλό να πάει κανείς με ένα αυτοκίνητο στον δρόμο και να μετρήσει εκεί τις ε, εκπομπές, αυτό φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν εξασφαλίζει την ε, ανθεκτικότητα, τη συγκρισιμότητα και την επαναληψιμότητα αυτών των δοκιμασιών. Θέλουμε ένα τεστ το οποίο να είναι πραγματικά αξιόπιστο και έχουμε δύο δυνατότητες σε σχέση με τα τεστ. Είχαμε δύο δυνατότητες και με τους εμπειρογνώμενους από τα κοινά κέντρα ερευνών είχαμε αναπτύξει αυτές τις δύο δοκιμασίες και φυσικά μετά από σύγκριση αυτό το τεστ το οποίο κρατήθηκε ήταν το καλύτερο αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή. Οι έρευνες αυτές βέβαια ήταν έρευνες σε βάθος. Όταν φτάσαμε στο τεστ αυτό, κάναμε και μία ψηφοφορία στην Τεχνική Επιτροπή για το τεστ αυτό τον προηγούμενο Μάιο. Δεν χάσαμε καθόλου χρόνο λοιπόν να αντιδράσουμε. Και τώρα, η πρόταση της Τι βρίσκεται στο τραπέζι των... Δεν είναι πρόταση. Όχι, είναι έγγραφα συζήτησης. Θέλαμε να έχουμε έγγραφα συζήτηση και να έχουμε και κάποια ανάδραση από τα κάτι μελη Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Σα λέω και πάλι, καμία πρόταση δεν έχει υποβάλει η Κομισιόν. Έχουμε ψήγματα προτάσεων βέβαια, γιατί πρέπει να συζητήσουμε με τα κάτι μελη Τι προβλέπουμε. Προβλέπουμε μια διαδικασία δύο σταδίων. Καταρχήν, θα τροποποιήσουμε τις, τους κανόνες για την ταχύτητα. Θα φτάνει μέχρι 160 χιλιόμετρα την ώρα με μέγιστο υψόμετρο 1200 μέτρα. Προβλέπουμε λοιπόν μια προσέγγιση σε δύο στάδια. Καταρχήν, από το 2017 να έχει γίνει το τεστ αυτό υποχρεωτικό. Από το 2016 θα εισαχθεί για λόγους ε, παρακολούθησης και υποπτήρες αλλά το 2017 θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αντανακλά αυτό το οποίο συζητήθηκε και στην ανακοίνωση CARS 2020 και στο δεύτερο στάδιο θα υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με, τον, με το όριο που θέτει ο κανονισμός αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το στατιστικό σφάλμα, δεν είναι κανείς τα 1000-1200 μέτρα κτλ. Δύο χρόνια αργότερα θα υπάρχει η πλήρης εφαρμογή. ο συντελεστής συμμόρφωσης. Αυτό είναι ένας παράγων ο οποίος μας επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις, ε, ε τις αβεβαιότητες που θα προκύψουν με την διαδικασία φορητών μετρητών εκπομπών και αυτός ο παράγων φυσικά θα συρρυκνωθεί προϊόντος του χρόνου. Επίσης η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή, για την έγκριση αυτή του κανονισμού είπαμε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε σαν στόχο στις 28 Οκτωβρίου να καταθέσουμε μια πρόταση. Γιατί θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα. Αυτό μας ζητήσανε κιόλα. Ο επόπτης ρυθμιστής. Σας είπα, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση, να συντονίσουμε τις ενέργειες των κρατών μελών τόσο διερευνητικά όσο και διορθωτικά να φτιάξουμε ένα σωστό τεστ για την, τις μετρήσεις και να εγκρίνουμε το σύστημά μας και για την έγκριση, να ενισχύσουμε το σύστημά μας για την έγκριση και για την εποπτεία. Έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε για όλα αυτά τα πράγματα, μετά από τα πρόσφατα αυτά γεγονότα. Αλλά τα γεγονότα αυτά μας οδηγούν να επανεξετάσουμε το αν αυτά που έχουμε είναι επαρκή, αν πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Όλα αυτά λοιπόν που είπατε είναι καλόδεκτα, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε μια τελική θέση. Περιμένουμε, προσπαθούμε να δούμε τις διάφορες ε, δυνατότητες και όλα αυτά τα οποία είχαμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή επανεξετάζονται στο φως των σύγχρονων των τελευταίων γεγονότων. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε τίποτα λοιπόν σε ό,τι αφορά την εξέβρεση μιας λύσης. Η προτεραιότητά μας είναι να δούμε τι έγινε και να προχωρήσουμε σε ένα πραγματικό τεστ το οποίο θα μετράει τις εκπομπές στο δρόμο, το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Κάποιοι θέλουν να επανέλθουν. Ο Ματίας Γκρότε πρώτα. Εντάξει. Εγώ είχα ζητήσει να μετριεται και η ποιότητα του αέρα, της ατμόσφαιρας σε ό,τι αφορά τα σωματίδια. Το πρόβλημα το βασικό είναι που έχουμε, προβλή, έχουμε κακή ποιότητα του, της ατμόσφαιρας της πόλης. Οι Βρυξέλλες δεν είναι στα 1200 μέτρα. Είναι ίσως στα 5 μέτρα ή κάτι τέτοιο. Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει 160 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να πιάσει κανείς τον αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία αλλά στις πόλεις, στι Βρυξέλλες, πού θα πάει κανείς με 160 την ώρα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση λοιπόν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα με το αν είναι κακή η ποιότητα της ατμόσφαιρας στις Βρυξέλλες. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι στα 95% των περιπτώσεων που δεν τρέχει κανείς με 160 την ώρα ή δεν είναι στα 1200 μέτρα θα είναι περιορισμένες οι εκπομπές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω από αυτά που μου λέτε. Πώς μπορώ εγώ να εξηγήσω σε ένα απλό άνθρωπο στην εκλογική μου περιφέρεια ότι κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τη ρήπανση του αέρα. Μου λέτε μετράμε στα 1200 μέτρα. Και όταν τρέχει το αυτοκίνητο με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι σχέση έχει αυτό με αυτό που γίνεται στις πόλεις. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα λοιπόν από αυτά που λέτε. Ήβο Μπέλετ, ένα σύντομο ερώτημα επίσης. Πρόεδρε, θέλω, λέει ο κύριος Μπελέτ, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτό το type approval, η ενίσχυση επίσης του ελέγχου στην αγορά, από αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι κάθε πληροφορία, κάθε input είναι ευπρόσδεκτο. Ναι, αλλά λέει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κάποια κεντρική υπηρεσία, περιμένει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι προς το παρόν είναι ε, η Εθνική Αρχή η οποία κάνει τους έλεγχους, αλλά εγώ νομίζω ότι αν θέλουμε να το αλλάξουμε, αύριο μπορούμε να έχουμε τη νέα πρόταση. Έχοντας και τα υπόλοιπα στοιχεία για το 2016 και 2017, μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα πολύ γρήγορα. Ήβο, σε ευχαριστούμε. Χέρμπραντι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και του εκπροσώπου τη Επιτροπή για τι απαντήσει του. Εκπροσωπείτε την Γενική Διεύθυνση που έχει την κυρίω αρμοδιότητα για την ανταγωνιστικότητα τη ε, βιομηχανία. Δεν έχετε την κυρία αρμοδιότητα για την ποιότητα ε, του αέρα της ατμόσφαιρας και γι' αυτό ακριβώς και εγώ θέλω να εστιάσω αυτό που σας λέω περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα γιατί προβληματίζομαι πάρα πολύ βαθιά για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε αλλά επίσης και για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διότι αυτή η περίπτωση της απάντησης από πλευράς Volkswagen είναι ένα αράπισμα τεράστιο για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γι' αυτό σας λέω, για άλλη μια φορά, παρακαλώ, να αλλάξετε την πολιτική σας για την διαφάνεια. Νομίζω ότι είναι πολύ απαράδεκτο, ιδίω σε μια τέτοια συγκυρία που τα διαβάζουμε όλα στις εφημερίδες κάθε μέρα. Ανοίγω την εφημερίδα και διαβάζω για κάποια έγγραφα τα οποία επισήμως ουδέποτε έχω λάβει και τα οποία τα έχετε εσείς στο σιρτάρι σας, τα έχουν και τα κράτη-μέλη στο σιρτάρι τους και συζητάτε τα της ε, συμμόρφωσης των συντηρητών συμμόρφωσης και έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι κάποια πρόταση. Μπορεί να πείτε ότι είναι θέμα διατύπωσης λέξεων, αλλά κυρίως είναι θέμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μια που δεν υπάρχει τέτοια, δεν υπάρχει διαφάνεια, ε, υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό σας λέω. Εκβάθρον να αλλάξετε την πολιτική σας για τη διαφάνεια και παρακαλώ να ε, προβείτε σε δημοσιοποίηση αυτών των ε, εγγράφων. Ε, όπως έχουμε και εμείς το δικαίωμα, έχουν δικαίωμα και οι Ευρωπαίοι να μάθουν τι συμβαίνει. Ε, Eichhout. Πρώτα-πρώτα να σα πω ότι είναι θετικό ότι τουλάχιστον ε, εγγράφο λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μας. Ε, αυτό είναι καλό και όπω λέτε εσεί υπάρχουν αυτά όλα γραμμένα, επομένω υπάρχει πρόταση. Οπότε, παρακαλώ, πέστε μας γιατί δεν δίνετε τις πληροφορίες σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα έγγραφα που υπάρχουν δεν τα κοινοποιείτε σε εμάς, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει κάποια διοργανική συμφωνία που ορίζει ότι θα πρέπει να είναι μια συμπεριφορά προς Συμβούλιο και προς Κοινοβούλιο. Να, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και κατά δεύτερον θέλω ακόμα να ξέρω τι λέει η νομική γνωμοδότηση, πώς μπορεί να αλλάξει το, το επίπεδο ενό κανονισμού μέσω της επιτροπολογίας γιατί αυτό κάνετε και με αυτό τον συντελεστή συμμόρφωσης το αλλάζετε, το αλλάζετε με τον κανονισμό αυτό από ό,τι ξέρω δεν προβλέπεται, δεν επιτρέπεται οπότε για πέστε μας ε, υπάρχει κάποια στατιστική ε, που το δικαιολογεί αυτό πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση για τις εκπομπές πραγματικής οδήγησης τότε θα προκύψει κάτι συγκεκριμένο και είπαμε για 43 μιλιγκράμμ ανά που είναι τα πρότυπα τα αμερικανικά άρα επ' αυτού θα πρέπει να ενεργήσετε και γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε αποκλίνει ο πρόεδρος και πάλι της κοιτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευχαριστώ Πρόεδρε τώρα. Για το πρώτο που ρωτήθηκε, ίσως δεν ήμουν σαφή, ίσως υπάρχει κάποια παρεξήγηση όταν είπα για τα 160 χιλιόμετρα και τα χίλια τα χίλια χιλιοστά ύψους. Ναι, ναι, για κάθε πόλη έχει άλλα, άλλες μεταβλητές, οπότε αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε με το φάσμα των τιμών. Το δεύτερο στοιχείο τώρα. Για την εποπτική ρυθμιστική αρχή. Τώρα μελετούμε όλα τα σενάρια. Πολλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά επίσης και η προηγουμένη εμπειρία και το τι γίνεται στην αγορά αλλά και το τι γίνεται σε σχέση με το πώς είναι οργανωμένοι άλλοι κλάδοι και τομείς. Τώρα, για τον συντελεστή συμμόρφωσης. Θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφές. Είναι και θέμα εμπειρίας η έγκριση της μεθοδολογίας των δοκιμών. Ξαρτάται βέβαια και από την κάθε δοκιμή να ποιος είναι ο ρόλος του συντελεστή συμμόρφωσης. Και βέβαια διαχρονικά είπαμε ότι σε δύο χρόνια θα υπάρχει πλήρες υλοποίηση. Οπότε με την πρώτη του χρόνου έχουμε περισσότερη εμπειρία για τα έγγραφα για την πρόταση. Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε κάποια έγγραφα εργασία, συζήτησης, επιλογές, πέστε το όπω θέλετε, εναλλακτικέ. Δεν υπάρχει κάποια αποκρισταλωμένη πολιτική της Κομισιόν τη Γενικής διεύθυνση. Κάνουμε ό,τι προβλέπεται στην Επιτροπή. Δεν έχουμε στη δική μα Γενική Διεύθυνση δικού μα κανόνε. Δεν ξέρω μήπως ο συνέλεφο θέλει να με συμπληρώσει. Ο άλλος κύριος είναι σημαντικό να μην παραμορφώνουμε τα περιστατικά και τα στοιχεία. Δεν έχουμε διαφορετικούς κανόνες. Έχουμε τη συνήθεια επιτροπολογία. Ακριβώς όπως υπενθυμίσατε, έχουμε ένα σχέδιο πρότασης για την εφαρμοστική πράξη που, που κοινοποιείται στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο. Και όπως σας είπε επανειλημμένος συνάδελφος, δεν υπάρχει στο τραπέζι κάποια πρόταση. Έχουμε κάποια τεχνοκρατικά, τεχνικά έγγραφα για κάποιες εναλλακτικές ε, που τα συζητούμε με τα κράτη-μέλη. Προχωράμε πολύ γρήγορα και μόλις τοποθετηθούν τα κράτη-μέλη για αυτές μας, για αυτά τα, τα στοιχεία, για αυτές, για αυτές τις εναλλακτικές, ε, τότε αμέσως πρόκειται να σας τα γνωστοποιήσουμε. σαν πρόταση. Και εσείς τότε θα ασκήσετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λυπούμε ε, για την κατάσταση, αλλά έτσι προβλέπεται. Έτσι ορίζει ο κανονισμός της επιτροπολογίας. Τα κάνουμε κάθε μήνα, τόσες φορές. Θα την πείτε, δεν διαφορετικό. Ο πρόεδρος. Συνάδελφοι, συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε τώρα κοινή συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή Ανάπτυξης και προηγουμένως έχουμε ένα ακόμα θέμα. Στις 5.30 είναι η κοινή συνεδρίαση. Το Κοινοβούλιο, όπως καταλάβατε, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τις απαντήσεις σας. Και μπορούμε εδώ να πούμε ότι ήδη σας προσκαλούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 9 Νοεμβρίου, 9 και 10 Νοεμβρίου. Να έρθετε και να μας εξηγήσετε την πρόταση. Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και εμείς θέλουμε να είμαστε καλά ενημερωμένοι για την πρόταση. Περιμένουμε λοιπόν τις εξηγήσεις σας για την πρόταση αυτή. Καλώς, οπότε τελειώνουμε με αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε στείλει κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω, συνεπώς, ότι μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρώτη ερώτηση. Και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με τις άλλες ερωτήσεις. Κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται πλήρως με το θέμα αυτό, παρακαλώ να μην μας ενοχλούν όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις ε, συζητήσεις τους για το προηγούμενο θέμα να τις συνεχίσουν εκτός αθούσης. Η Μαριάν Βένιγκ έχει τώρα το λόγο λοιπόν που είναι διευθύντρια για την ποιότητα ζωής, ε, τα ύδατα και τον αέρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Για την πρώτη ερώτηση, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δύο γύρους αξιολόγησης. Έγινε μια πρώτη έκθεση το 2012 και μια δεύτερη το 2014. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις χώρες μέλη θα πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που αναφέρονται στην οδηγία για τα ύδατα. Έχουμε αναγνωρίσει λοιπόν τις προσπάθειες που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη προκειμένου να πετύχουν ε, τους στόχους αυτούς και έχουμε μερικά πολύ καλά παραδείγματα και επιτεύγματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι η βάση των όσων σήμερα γνωρίζουμε, ο στόχος του 2015 για καλή ποιότητα ε, ύδατος δεν έχει επιτευχθεί. Τι κάνουμε λοιπόν. Πιστεύουμε ότι οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα. Αυτό είναι πολύ βασικό να το λάβουμε υπόψη μας στο δεύτερο στάδιο των διαχειριστικών σχεδίων που θα μας υποβληθούν τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς. Σε ποιους τομείς είναι σημαντική βελτίωση. Περιμένουμε να κάνουν βελτίωση στον έλεγχο οι χώρες μέλη, στην αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων και της ποιότητάς τους. Επίσης θέλουμε να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα και θα επανέλθουμε γι' αυτό για την ε, ρήπανση η οποία διαχέεται στο είδωρ και που προκαλείται από την γεωργία. Τα μέτρα λοιπόν πρέπει να ξεφύγουν ε, από την πεπατημένη και να δούμε και την γεωργική πολιτική για να βελτιωθεί η κατάσταση των δάτων. Το τρίτο που θέλουμε να κάνουν οι χώρες μέλη είναι τα εδάτινα σώματα τα οποία πλήττονται από αλλαγές στη ροή στο σχήμα θα πρέπει να κοινοποιούνται καλύτερα και οι χώρες μέλη θα πρέπει να παίρνουν ό,τι μέτρα χρειάζεται και να μας εξηγούν γιατί παίρνουν αυτά τα μέτρα και όχι άλλα. Είναι κάτι το οποίο δεν το είδαμε στα πρώτα σχέδια διαχείρισης των ε, υπογειών υδάτων των λεκανών και θα έπρεπε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν σιγά σιγά οι αρνητικέ επιπτώσεις που έχουν να κάνουν ναι, με την αλλαγή στη μορφολογία. Και το τέταρτο που περιμένουμε από τις χώρες μέλη είναι ότι πιστεύουμε πως οι χώρες μέλη δεν συμμορφώνονται με τον καλύτερο τρόπο στην αρχή της ε, ανάκτησης του κόστους προκειμένου να δοθούν κίνητρα ώστε να καθαρίζονται οι περιοχές εκείνες που υποφέρουν από ρήπανση των υδάτων. Οι χώρες μέλη δεν παίρνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να υπογραμμίσω και δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι και εσείς είχατε μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας ε, για τα ύδατα με 8 δισεκατομμύρια το χρόνο αλλά αυτά πάνε χαμένα αν δεν έχουμε σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Και νομίζω ότι σας δώσαμε την στήριξη που θέλατε προκειμένου να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και προκειμένου να έχουμε αυτά τα ωφέλη. Χτες ήταν εδώ ο Γενικός μου Διευθυντής, ο οποίος μίλησε για την ε, μεσοπρόθεσμη έκθεση όσον αφορά την βιοπικιλότητα. Και είπε ότι και το είδωρ αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα και η καλή κατάσταση όλων των υδάτινων σωμάτων για να επιτευχθούν ακριβώς και αυτοί οι στόχοι της βιοπικιλότητας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο εισηγητής, ο κύριος Γκάμπους, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για το θέμα των υδάτινων χώρων στα κράτη-μέλη. Λέει η Κομισιόν στο έγγραφό τη για την οδηγία για το είδαρ και τι ε, πλημμύρε ότι πολλά κράτη αναρωτήθηκαν πώ μπορεί κανεί να προχωρεί για τα θέματα αυτά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε είδωρ στα σχέδιά τους, κάτι το οποίο τους υποχρεώνει η οδηγία πλαίσιο για, το, για, τα, για τους υδάτινους πόρους. Υπάρχουν πολύ, πολλά κακά παραδείγματα. Η λεκάνη του Εύρου, παραδείγματο χάρη του Ισπανικού Εύρου, έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τις υδάτινες μάζες, όπως λέει η Κομισιόν. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι πληροφορίε συμπληρωματικέ που δόθηκαν από την Ισπανική κυβέρνηση μετά από την ολέθρια έκθεση τη Κομισιόν που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο θεωρείται και πάλι ότι καλύπτουν την οδηγία πλαίσιο. Τον Απρίλιο, σε απάντηση σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση, είπε η Κομισιόν ότι τα προγράμματα για τις ε, ισπανικές υδρογραφικές λεκάνες πιο αργά, του λέει ο πρόεδρος. Σε παρακαλώ. Τον Απρίλιο, λοιπόν, στην απάντηση σε μια ερώτηση, είπε η Κομισιόν ότι τα προγράμματα για τις υδρογραφικές λεκάνες της ε, Ισπανίας και η ροή, η παροχή των ποταμών δεν είναι σαφές ότι καλύπτουν τα οικολογικά σχέδια. Στο σχέδιο λοιπόν για τον Εύρο το 2015-2016 δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ του σχεδίου 2009-2015 που ενεκρίθηκε το 2014. Το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν βρίσκεται στην καθυστέρηση για την εκπόνηση των σχεδίων από την προηγούμενη σοσιαστική κυβέρνηση. Η κατάσταση όμως των υδατίνων πόρων σε ένα κράτος μέλος σε, δεν μπορεί να οφείλεται σε κακή διαχείριση όπως συνέβη σε αυτήν την περίπτωση. Γι' αυτό ήθελα να ζητήσω από την Κομισία μας ποια είναι η άποψή σου για τα σχέδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί και αν έτσι όπως έχουν διατυπωθεί μπορούν να εξασφαλίσουν το σεβασμό των οικολογικών στόχων και τις απαραίτητες παροχές ύδατος που προβλέπονται από το, από σχέδιο για τους υδάτινους πόρους. Ευχαριστώ. Κυρία Σογκέρ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι με αυτή την ερώτηση. Την ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Γεωργία, γιατί συζητάμε στην Ολλανδία πάρα πολύ για τα φωσφορικά. Για τα 50 mg. τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους δείκτες δηλαδή και για τα όρια που έχουμε βάλει. Πρόκειται για καθαρά ύδατα. Ο καθένας όμως βλέπει διαφορετικά τις προδιαγραφές. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θέλω την έκθεση που λέει ότι η Γεωργία είναι υπεύθυνη για το 90%. Όμως οι διάφοροι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη σας και τις αποχετεύσεις και όχι μόνο τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει τώρα το λόγο. Εγώ χαίρομαι πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε έστω σύντομα για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που βέβαια είναι η διαχείριση των υδάτων σε όλες τις μορφές. Και εκεί λυπούμε να πω ότι η έκθεση που ειδικά αφορά την Ελλάδα αντανακλά μια αντιμετώπιση του θέματος από την ίδια την ελληνική πολιτεία γεμάτη με καθυστερήσεις, ελλείψεις και παραλήψεις. Δεν ξέρω, στην καλύτερη περίπτωση αυτό δείχνει διοικητική αδυναμία και στη χειρότερη όμως πολιτική αδιαφορία για την εφαρμογή της οδηγίας. Θέλω να τονίσω από την άλλη μεριά ότι ο ελληνικός λαός αγαπά και ενδιαφέρεται για το πλούσιο, το εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον της χώρας και θεωρεί την προστασία του σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι αποτελεί προτεραιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω ορισμένες, αν μου επιτρέπετε, σχετικές ερωτήσεις σε ποιο βαθμό έχει αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εργαλεία τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο. Τι, δεύτερη ερώτηση, τι μπορεί πραγματικά, ρεαλιστικά να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εδώ και πέρα ώστε να ασκηθεί πίεση αλλά και να δοθούν ίσως κίνητρα ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος ε, ίσως γνωρίζετε ότι ο πρώτος κύκλος των ενεργειών έχει περίπου χαθεί ήδη. Και τελευταία ερώτηση, τι πρέπει να κάνει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, η καινούργια ελληνική κυβέρνηση σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο, ώστε να μπει σε τροχιά εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Ε, εν κατακλείδη Πολλές φορές έχω παρατηρήσει κύριε Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αρέσκεται στα μεγάλα λόγια αλλά η απόσταση μέχρι την πράξη στα επιμέρους κράτη είναι πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε πολύ μεγάλη. Πρέπει να μάθουμε, αυτό είναι ίσως το δίδαγμα για μένα, την απόσταση αυτή να τη μικρύνουμε όσο μπορούμε και μια θεωρία να ακολουθεί γρήγορα η οδηγία και η πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναγυρίζω στην Κομισιόν για τις απαντήσεις που πρέπει να μας δώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν για το αν επιτυγχάνουμε πρόοδο στην έγκριση του δευτέρου, το, της δεύτερης φάσης για τα σχέδια διαχείρισης υδατίνων λεκανών, λεκανών ποταμών συγκεκριμένα. Εμείς συνεχίζουμε τις επαφές με τα κρατημέλη για να εξασφαλίσουμε ότι ακολουθούν τη διαδικασία με τις δημόσιες διαβουλεύσεις, γιατί όλα αυτά πρέπει να περατωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Και όπως είπα προηγουμένως, το Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να υποβληθούν όλα αυτά τα στοιχεία στην Κομισιόν. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις στον πρώτο γύρο και αυτό ήταν λυπηρό. Και υπήρξαν και ορισμένες δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με τις καθυστερήσεις αυτές, αλλά προσπαθούμε καταρχήν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και με διμέρειες επαφές προσπαθούμε να τους πείσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και προσπαθούμε να υποδείξουμε και τα σημεία όπου υπάρχουν πραγματικά <coughs> μη ικανοποιητικέ διατάξεις στα πρώτα του σχέδια για τη διαχείριση ποταμίων λεκανών. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ως προκατακτικές αξιολογήσεις για το δεύτερο σχέδιο που θα υποβάλει το κάτι μελη Μπορούμε λοιπόν να ελπίσουμε ότι στο δεύτερο γύρο θα έχουμε καλύτερη πληροφόρηση όχι μόνο για την κατάσταση των λεκανών των ποταμών αλλά και για την παρακολούθηση, τα μέτρα παρακολούθησης και τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσουν για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις. Για την οδηγία περινητρικών αλάτων υπάρχει το όριο 15 μικρογράμμ το, στο λίτρο. Αυτό είναι μια σταθερή τιμή στην οδηγία για τα νητρικά άλατα. Αυτό βέβαια δεν εξασφαλίζει την υγεία του οικοσυστήματος, εξαρτάται από το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά φυσικά η οδηγία ξεπερνάει την ε, οδηγία μόνο για τα νητρικά άλατα σε ό,τι αφορά την ε, επίτευξη του οικολογικού αυτού επίπεδου <clears throat> ποιότητος. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε ένα από τα μεταγενέστερα ερωτήματα που θα διαλάβω. Ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι εδώ. Να πω κάτι για την γεωργία και τους σωλήνες ε, που έχουν διαρροές. Έχουμε σημειακές πηγές και διάχυτες πηγές ε, ρήπανσης. Δεν λέω ότι οι σημειακές πηγές δεν συμβάλλουν και αυτές στο γεγονός ότι δεν έχουμε ικανοποιητικό καθεστώς περιβάλλοντος. Ξέρουμε όμως ότι οι διάχυτες πηγές ρήπανσης είναι οι πιο ουσιαστικές και γι' αυτό ανέφερα αυτά τα στοιχεία που είπα για τον αντίκτυπο από την γεωργία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Thank you very much. Now we can... Ευχαριστώ και πάλι. Τώρα μπορούμε... Ναι, για αυτό το σημείο θέλετε να το λόγο. Μετά. Εντάξει. Έχουμε ένα άλλο σημείο μετά, ναι. Δεύτερο ερώτημα τώρα και ζητώ από την Κομισιόν να δώσει την απάντηση για το δεύτερο σημείο και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτό το δεύτερο σημείο. Όσο προχωράει η συζήτηση, απαντάμε και στις άλλες ερωτήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εφαρμόσουμε καλά την οδηγία. Το 2015, όπως είπα και πριν, τέθηκε χρονικό όριο για να πετύχουμε την ε, καλή κατάσταση των υδάτων. Δεν το πετύχαμε. Κατά 53% χώρες μέλη το έχουμε πετύχει. Α, 53% των υδάτινων σωμάτων. Πρόκειται για βελτίωση όμως θα έλεγα γιατί αν το συγκρίνουμε το 2009 υπάρχει βελτίωση 10%. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε 10.000 επιπλέον υδάτινα σώματα τα οποία βρισκόνται σε ανάκαμψη. Τώρα εξαρτάται αν κανείς βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Πάντως θέλω να κάνω μια παρατήρηση γιατί ναι, δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει πρόοδος με τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται, όχι βέβαια αμέσως όχι μέσα στην ίδια χρονιά ή μέσα στην επόμενη. Χρειάζονται πολλά χρόνια για να βελτιωθεί η κατάσταση, να μειωθεί δηλαδή η ρήπανση και να έχουμε τους στόχους που θέλουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τίποτα δεν πάει καλά. Ναι. Αντίθετα, με την βελτίωση βελτίωση στην οποία μόλις αναφέρθηκα πιστεύουμε ότι η τάση είναι θετική και ελπίζουμε ότι θα δούμε την ίδια τάση να επιβεβαιώνεται και με τα νέα δεδομένα που μας έρχονται από τις χώρες ε, μέλη όταν θα μας στείλουν δηλαδή τις εκθέσεις τους για την ε, διαχείριση των υδάτρων λεκανών. Τώρα, κατά τα άλλα σας είπα ότι έχουμε συμπληρωματικέ δράσεις και με άλλες ε, οδηγίες, με τα νητρικά, χημικά και άλλη νομοθεσία δηλαδή και θα συνεχίσουμε και πάλι όπως είπα και το επαναλαμβάνω ότι έχουμε στενές επαφέ με τις χώρες μέλη. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία στρατηγική εφαρμογής Οπότε είτε πρόκειται για τη γεωργία, είτε πρόκειται για οικονομικά, είτε πρόκειται για ανταλλαγή δεδομένων. Τα συζητάμε με τις χώρες μέλη και προσπαθούμε να βρούμε κοινό τόπο. Μια ενιαία δηλαδή ερμηνεία για την οδηγία για τα ύδατα, οπότε από εκεί και πέρα οι χώρες μέλη μπορούν να προχωρήσουν σωστά. Βέβαια, αν τα μηνύματα δεν περνάνε, ε, προχωρούμε σε δράση επιβολής, συμμόρφωσης. Πηγαίνουμε δηλαδή στην ε, διαδικασία επιπαραβάση. παραβάση, τη δικαστική διαδικασία. Και βλέπουμε αν ε, λύνονται τα προβλήματα στο μεταξύ ή όντω θα ε, δικαστούν στο δικαστήριο. Τώρα μια άλλη πτυχή, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα, είναι η οικονομική στήριξη που διατίθεται μέσω των διαφόρων εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα, το Περιφερειακό και Αναπτυξιακό Ταμείο και που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα χώρη μέλη. Μερικές φορές υπάρχει το Γεωργικό Ταμείο παρεμβαίνει και δεν χρησιμοποιούνται πάντα ε, τα κονδύλια για το σκοπό που προβλέπονται. Τέλος, βασιζόμαστε πάρα πολύ στη δικιά σας στήριξη. Στις χώρες σας δηλαδή, προκειμένου να μας βοηθήσετε και μας. Η... Το σχέδιο αυτό διαχείρισης να προχωρήσει, να τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρηθούν και τα κράτη-μέλη να ενισχύουν τις προσπάθειές τους, όχι μόνο να μας στέλνουν τις εκθέσεις τους έγκαιρα, αλλά να υιοθετούν και τα σωστά μέτρα πολιτικής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Eckhout. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα και επί τη βάση των ερωτήσεων που τέθηκαν, βλέπω ότι υπάρχει μια θετική τάση. Αλλά υποτίθεται ότι το 2015 τα πράγματα θα ήταν όλα εντάξει. Καλό είναι να υπάρχει σωστή πορεία, αλλά αν έχετε μονάχα βελτίωση 10% σε 5 χρόνια, αυτό είναι πολύ χαμηλή βελτίωση. Δεν νομίζω ότι το ΕΚΟΦΗΝ θα ήταν ικανοποιημένο με μια τέτοια βελτίωση της τάξης του 10%. Άλλοι κανόνες φαίνεται ότι εφαρμόζονται εκεί. Και τώρα, πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την ανακοίνωση που είπατε για την εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα. Ξέρετε ότι πολλά κράτη-μέλη το απλώς ακολουθούν αυτό το οποίο θα κάνανε ούτως ή άλλως, business as usual και λέτε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπαθίες μου. Εγώ δεν ξέρω όμως πότε η Κομισιόν θα αρχίσει να σκληρέ λιγάκι τη στάση της για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα αυξήσουν τις προσπαθίες τους. Γιατί βλέπουμε ότι για πολλά κράτη-μέλη δεν γίνεται καμία πρόσθετη προσπάθεια. Επικοινωνούν μαζί σας, λένε ότι είναι έτοιμα να δράσουν, δεν κάνουν τίποτα για να αναβαθμίσουν τις προσπαθίες τους. Μήπω μπορείτε να είστε λίγο πιο επακριβείς. Λέτε θεωρητικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλα μέτρα ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά είναι βέβαια το οπλοστάσιο που έχετε στην, ε, στη διάθεσή σα. Αλλά τι θα κάνετε τελικά αν ένα κράτος μέλος δεν βελτιώσει τι προσπάθειέ του. Πότε εσεί θα εξασφαλίσετε ότι κάνει κάτι περισσότερο. Θα το κάνετε στο τέλος του 2015 αν δεν το κάνει τώρα στο 2015, πότε θα αναλάβετε δράση. Θέλω να έχω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι να μας εξηγείτε ποιο είναι το γενικό πλωστάσιο που έχει στη διάθεσή σας και το τι θα μπορούσατε δυνητικά να κάνετε. Είναι καιρό, καιρός η Κομισιόν να είναι λίγο πιο αυστηρή όπως είναι και οι αντίστοιχε διευθύνσεις στα οικονομικά για τα οικονομικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, και δεν βλέπω, δεν είμαι βλέπων άλλους συναδέλφους που να θέλουν να λάβουν το λόγο συγγνώμη. Ε, θα συνεχίσω στο ίδιο ύφο με τον προηγούμενο συνάδελφο και εγώ μίλησα ειδικά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Πήρα γενικές διαβεβαιώσεις για όλα τα κράτη, αλλά τίποτα πιο συγκεκριμένο. Και το 53% που ανέφερε η κυρία ε, της ε, Κομισιόν είναι δύσκολο να τα ορίσω αν είναι οπισθοχώρηση ή πραγματική πρόοδος. Νομίζω ότι επαναλαμβάνω το θέμα των υδάτων είναι εξαιρετικά σοβαρό και για το λαϊκό κόσμο και για μας τους ευρωβουλευτές και πρέπει επιτέλους να δούμε πιο συγκεκριμένη πρόοδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, uh, Miss ευχαριστώ πολύ και την λόγω στην κυρία Ντέλη. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με κράτη-μέλη που ίσως ισχυριστούν ότι υπάρχουν επιπλέον προβλήματα όσον αφορά τη βελτίωση του, του αέρα και των υδάτων σε σχέση με τους υδάτινους πόρους και τι θα γίνει. Πώς θα εξασφαλίσετε αυτή τη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας θα ολοκληρωθεί σε εκείνες τις χώρες. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα ληφθούν υπόψη αυτές οι επιπλέον προκλήσεις. Ο πρόεδρος στο πάρα πολύ και δίνει το λόγο στην κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι εδώ εξ του κύριου Γιάννου Βίτεμα, του συναδέλφου μου, ο οποίος έχει θέσει δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Είναι οι ερωτήσεις 4 και 8 αν δεν κάνω λάθος, θα ήθελε η Κομισιόν να της απαντήσει ή δυνατόν. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω, δεν τις έχω μπροστά μου, αλλά νομίζω η Κομισιόν τις έχει. Εμείς λειτουργούμε έτσι, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Ε, έτσι, έτσι, το, έτσι το κάνουμε. Ξεκινούμε μια πρώτη ερώτηση, κατόπιν ε, απαντάτε και κατόπιν ξεκινούμε μια άλλη ερώτηση. Αλλά θα μπορούσατε να περιμένετε και θα ακούγατε την ερώτηση. Την απάντηση, συγγνώμη. Και τώρα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Α, όχι, συμπαθάτε με κύριε Πελίτσιν, Μόνο ένα πραγματάκι να προσθέσω σε σχέση με όσο είπε ο κύριο Μπάς Έκχαουτ. Εμείς καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα. Μας και αυτό στην Ιταλία. Υπάρχει ένα μέρος που αντάγριο ονομάζεται που έχουμε καταστάσεις ε, πετρελαϊκές και από εκεί περνάει επίσης το πόσιμο είδωρ για βασιλικά τα ε, Καλαβρία ή όλο το νότο της Ιταλίας και τελικά αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει ε, ρήπανση από τους υδρογονάνθρακες ε, και από διάφορα βαρέα μέταλλα οπότε όλα αυτά τα καταγγείλαμε στην Κομισιόν η οποία ξεκίνησε μία διαδικασία επί πέρασε ένας χρόνος, ε, δεν έγινε τίποτα. Ακριβώς όπως είπε ο κ. τι γίνεται, άπαξ και φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο, εσείς έχετε ενημέρωση για αυτό το οποίο γίνεται, γιατί έχουμε παραβίαση σημαντικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων, δηλαδή το δικαίωμα στην υγεία. Τι πρέπει να κάνετε, τι κάνετε για να προστατεύσετε την υγεία του κόσμου, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη ερώτηση. Εάν δεν έχουμε να λάβει το λόγο η Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για πολλά θέματα και εσείς έχετε υπογραμμίσει αυτό το θέμα αλλά ισχύει και για το ερώτημα που μόλις ετέθη Αυτά για μένα συνδέονται με το ερώτημα υπαριθμών 8, στο οποίο θα απαντήσω αργότερα, αν μου επιτρέπετε. Για το τι κάνουμε και πώς εμείς θα προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα βήματα. Όπως είπα, κάνουμε δύο πράγματα, έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μιλάμε πολύ και πολύ εντατικά με τα κράτη-μέλη για να τους επιτρέψουμε να καταλάβουν να φτάσουν σε μια κοινή συναντήληψη για το πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Θεωρούμε ότι αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχουμε εξασφαλίσει μια μεγάλη πρόοδο στην ε, εφαρμογή. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που ήμασταν, δεν είχαμε αυτή τη διαδικασία συνεννόηση με τα κράτη-μέλη. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, είναι εντατικοποιούμενη, αλλά Έχουμε και τις διαδικασίες επί παραβάση. Αν δείτε τον τομέα των υδάτων έχουμε περίπου 30 με 40 διαδικασίες επί παραβάση. Όχι μόνο αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία για τα, τους υδάτινους πόρους, αλλά και για τον, τους οντροφόρους ορίζοντες, το νερό στις πόλεις κτλ. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάσεων. Το είδωρο είναι ένας από τους τομείς όπου είναι πολλές αυτές οι διαδικασίες. Εμείς παρακολουθούμε όσο μπορούμε τις νομικές αυτές διαδικασίες, δικαστικές διαδικασίες, αλλά σε τελική ανάλυση α, είναι τα κάτι μέλη τα οποία θα πρέπει να δράσουμε. Και εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχει ο γενικός στόχος το 2015 να επιτύχουμε μια καλή κατάσταση του περιβάλλοντος. Θα θυμόσαστε όμως ότι στο αυτό Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Και αν χρησιμοποιηθούν αυτές οι εξαιρέσεις, μπορούμε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να φτάσουμε το 2027, πάντα με τις κατάλληλες δικαιολογίες. Και είχαμε πολλές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για το δεύτερο σχέδιο για τις υδάτινες λεκάνες ποταμών Εκεί οι προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις είναι πολύ πιο στεναρές από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Για την Ελλάδα τώρα. Το τελευταίο σχέδιο από την Ελλάδα που ενεκρίθη τον Αύγουστο του 2015 μόλις το πήραμε και το εξετάζουμε. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια αξιολόγηση, ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εν παραλίλω συζητάμε πάρα πολύ με την Ελλάδα για να υπάρξει πρόοδος για το δεύτερο σχέδιο για την, ε, τις λεκάνες ποταμών. Οπότε η ελλείψη του πρώτου σχεδίου να μην επαναληφθούν στο δεύτερο. Για την ε, λειψιδρία και το τι γίνεται τότε με την οδηγία πλαίσιο, φυσικά η οδηγία δεν αφορά μόνο την ποιότητα του ύδατος αλλά και την ποσότητα του ύδατος. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση ξηρασιών που τα, οι κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ελπίζω λοιπόν ότι έτσι έχω απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματά σας. Κάποια από αυτά βέβαια θα απαντηθούν στις ε, ε, επερχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πάμε στην τρίτη ερώτηση για τα σχέδια διαχείρισης υδάτων και πάλι δυνατό το λόγο στην Κομισία να Ευχαριστώ. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην οδηγία και την ερμηνεία τους. Θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η απόφαση λέει ότι όλα τα νέα προγράμματα δεν θα μπορούν να εγκριθούν ή να εφαρμοστούν. Εμείς ε, το βλέπουμε ως εξής. Επιβεβαιώνεται η γραμμή αντίστοιχων ρυθμίσεων που λένε βασικά ότι σκεφτείτε πριν δράσετε. Δηλαδή πρέπει να αξιολογήσετε τη δράση σας πριν προχωρήσετε για να υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα σε όλα όσα διακυδεύονται. Η αξιολόγηση τώρα πριν από την άδεια είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Υπάρχει και με την οδηγία ΙΕ και με την οδηγία για τους οικότοπους. Αν επιδεινώνεται ε, η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων πρέπει να καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις οδηγίες. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν αλλάξει μετά την απόφαση του δικαστηρίου και σχέδια που πρέπει να περάσουν από αντίτυπο επιπτώσεων ή από την οδηγία για τους οικότοπους Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή βάσει όλων αυτών, να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορούν να υπάρχουν νέα σχέδια εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Και ακόμα και αν τέτοια σχέδια καταλήγουν σε επιδείνωση των υδάτων βάσει της οδηγίας για τα ύδατα, μπορούν να προχωρήσουν αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις και τους όρους για τις εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 7. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή του σχεδίου, να τροποποιηθεί για να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία και το ότι δεν μπορούν ε, όλα τα σχέδια να προχωρήσουν όπως έχουν ε, αρχικά σχεδιαστεί αλλά πρέπει να τροποποιηθούν, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως αποδεκτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μισελ Νταντά. Ε, χωρίς μικρόφωνο όμως δεν τον ακούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επεξηγήσεις της. Η απόφαση του δικαστηρίου, στην οποία αναφέρεται, δείχνει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ερμηνεία μεταξύ των χωρών μελών για το θέμα αυτό ακριβώς της επιδίνωσης της κατάστασης των υδάτων και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύσουμε τα έργα τα οποία προτείνονται. Το παράδειγμα ε, πρόκειται για μια αλλαγή για οικονομικούς λόγους, για να μπορέσουν να περνάνε πιο μεγάλα πλοία. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει προσωρινά επιδείνωση με έργα τα οποία έχουν ως τελικό στόχο να βελτιώσουν την κατάσταση. Το πρώτο είναι εκείνο το, το Ρομοντάνιο, όπου έπρεπε να βγάλουμε χώμα για να μην κινδυνεύουμε από πλημμύρες. Υπάρχει μια επιδείνωση όσο προχωρούσε το εργοτάξιο, αλλά υπήρξε αποκατάσταση μετά. Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις πλημμύρες πάλι και είναι εκείνο των Μπέρς προκειμένου να εφαρμόσουμε πραγματικά μία οδηγία για να αποφύγουμε δυσκολίες ερμηνείες ανάμεσα στην οδηγία για τα ύδατα και την οδηγία για τις πλημμύρε. Ρωτάω λοιπόν, μεσοπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει ε, την ε, απόφαση έτσι ώστε να είναι πιο συγκεκριμένη και να μην επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες και να βελτιώνει πράγματι ε, μακροπρόθεσμα την ποιότητα των υδάτων και του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε για αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει Κανένα άλλο που θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. <coughs> Καλώς. Οπότε το λόγο έχει και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> <coughs> ναι. Μία διευκρίνηση που θα ήθελα να κάνω για την οδηγία, η οδηγία πλαίσιο του ύδατος δεν αφορά τις, ε, δεν ασχολείται με τις προσωρινές υποβαθμίσεις του περιβάλλοντος, όμως δεν υπάρχει καμία σύγκρουση εδώ. Το άλλο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω. Αυτά τα εφαρμόσουμε από το 2008. Έχουμε την κοινή στρατηγική <clears throat> εφαρμογή, είναι διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως και που αφορά και τις εξαιρέσεις και η απόφαση του δικαστηρίου συνάδει με αυτές τις κατευθύνσεις και τη γραμμή πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Κομισιόν η οποία έτσι επιβεβαιώνεται μέσω της δικαστικής απόφασης και έχουμε τώρα ένα πρόγραμμα εργασίας 2016-2018 συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και θα συζητήσουμε και πάλι αυτή τη δικαστική απόφαση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είναι συνεκτική η ερμηνεία που θα δοθεί σε αυτήν την απόφαση από τα κατημέλη, ότι την καταλάβαν τα κατημέλη θα την εφαρμόσουν με ομοιόμορφο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, λέω Μπορούμε τώρα να πάμε στο επόμενο ερώτημα, το σημείο συνδέσεις με άλλες περιοχές πολιτικής 4-4 ρήπανση που προέρχεται από την Γεωργία και δεν το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέχυψε και στο παρελθόν. Μπορώ να πω μονάχα είμαστε σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τα νητρικά άλατα αυτό δεν ε, είναι της άμεσης αρμοδιότητάς μου, αλλά φυσικά έχει επιπτώσει την οδηγία περί υδάτων και υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για την ε, εφαρμογή με την Επιτροπή Νητρικών Αλάτων που βοηθάει την Κομισιόν στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Υπάρχει βέβαια κενό στις ε, εφαρμογές σε πολλά σημεία και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την, τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ομοιόμορφη εφαρμογή, εν ανάγκη και με δικαστικές διαδικασίες και η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες επί παραβάση και επίσης με τα κράτη-μέλη που ετοιμάζουμε την εντολή για την κοινή στρατηγική εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα τα επόμενα δύο χρόνια και στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και τα θέματα τα οποία επηρεάζουν τον τομέα της γεωργίας και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στις συζητήσεις με τα κρατη για να έχουμε μια νέα ερμηνεία, να αναπτύξουμε κοινέ λύσεις, να αντιμετωπίσουμε τα πιο πιεστικά προβλήματα που έρχονται από την διάχυτη ρήπανση και από τις αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους. Στις διμερείς επαφές με τα κράτη-μέλη έχουμε αναφέρει ότι το κενό αυτό υπάρχει σε βασικά μέτρα και ότι θα χρειαστεί όχι μονάχα να εξετάσουμε την εφαρμογή των βασικών μέτρων αλλά θέλουμε να δούμε στον επόμενο γύρο των σχεδίων διαχείρισης υδατίνων λεκανών ποταμών να υπάρχει και η δυνατότητα ή ας το πω αλλιώς η ανάγκη για τα κατημέλη να προχωρήσουν επέκεινα των βασικών μέτρων. Και υπάρχει το θέμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένα θέμα περιλαμβάνεται στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά όχι στην οδηγία με τα, για τη βιώσιμη χρήση των ε, παρασιτοκτόνων και ζυζανιοκτόνων. Η Κομισιόν εργάζεται με τα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα στους ίδιους τους κόλπους, για να δει πώς η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί στο βαθμό του δυνατού, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και το θέμα αυτό της πολλαπλής συμμόρφωσης ό,τι αφορά το, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Μόλον τούτο υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί και μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουμε ότι ο αγροτικός τομέας έχει την δυνατότητα εκπλήρωσης ή αρρωγής της εκπλήρωσης αυτών που επιτάσσει η οδηγία για την ποιότητα των υδάτων υπάρχει η υποχρεωτική ε, δημιουργία ενός σώματος συμβουλευτικού για τους γεωργούς όπου οι γεωργοί έχουν όλοι το δικαίωμα πρόσβαση σε αυτό το φορέα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι συμβουλές για την εφαρμογή των μέτρων. Η πολιτική για την εκπόνηση κανόνων και αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο μέσω της νέας, ε, του νέου κανονισμού για την εξέλιξη των κανόνων και της ε, συναφούς νομοθεσίας είναι φανερό ότι μέσα στην ίδια την πυρηνική νομοθεσία, τον πύρινα της νομοθεσίας υπάρχει δυνατότητα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των, της των υδάτων και συγκεκριμένα στη γεωργία. Αυτό είναι μια επιταγή που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα κάτι μελη όταν δαπανούν μέσα στη διαδικασία εκπόνησης κανόνων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που είναι διαθέσιμο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτές τις προτεραιότητες, βοήθεια, συμβουλές ε, για πολιετή χρυσή γης, επενδύσεις, κατάρτιση κτλ. Με όλα αυτά τα μέλη μπορούν να προχωρήσουν. Το 2017 έως 2019 θα έχουμε τις αιτήσει εκθέσεις εφαρμογής που θα έρθουν από τις διαχειρίστριες αρχές των προγραμμάτων και τότε εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση των ε, κανόνων για την αγροτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα. Έχεις δει στο κυρία Ούκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα Δανέζικα. Ξέρετε, Πρώτα πρώτα. Πρέπει να σας πω ότι τώρα έχουμε αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι πολλά η πλειοψηφία των μέλων της Ένωσης δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Και να σας πω την ίδια μου τη χώρα, όπου η κυβέρνηση δεν έχει Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συγχωνεύτηκε με το Υπουργείο Γεωργίας. Το κατάπιε το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το πρώτο το οποίο έγινε είναι, ήταν η αναθεώρηση των θεσπιστέντων νόμων σε σχέση με κάποιες προστατευμένες ζώνες. Ας πούμε, ε, υπήρχαν κάποιο είδου ε, φράγματα για ε, τη ροή των υδάτων. Αυτά έχουν τεθεί ένα αμφιβαλό, οπότε βλέπετε τι κάνει η δανέζικη κυβέρνηση. Έχει λάβει υπόψη της αυτή την κατάσταση η Επιτροπή. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ στη Δανία. Ήταν γνωστό ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χώρα μου. Αλλά υποθέτω ότι είναι μόνο η Δανία. Θα γίνεται και σε άλλες χώρες, γιατί η Δανία άλλωστε ε, είναι η χώρα με τις πιο πυκνές, τις πιο πολλές καλλιέργειες. Οπότε πάρα πολύ δύσκολο κάτι να αλλάξει. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με ναι, όλες αυτές τις φήμες που λένε ότι υπάρχει υπερβολική, ακραία εφαρμογή ε, του δικαίου στην ε, Δανία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Ε, θα πρέπει να το προλάβει αυτό υπόψη και το ελεγκτικό συνέδριο γιατί έχει διατυπώσει κάποιες συστάσεις βελτίωση της κατάστασης ότι δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλα όσα έχουμε θεσπίσει για τις συνθήκες ε, άσκησης της γεωργίας θα πρέπει να τηρούνται όσο προβλέπονται. Βλέπουμε ότι έτσι αμφισβητούνται οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαμε αυτό γίνεται μόνο στην Δανία, γίνονται και αλλού. Οπότε θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας μέχρι ότου βελτιωθεί η κατάσταση. Και Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και στη χώρα μου αλλά και αλλού ε, έχουν μολυνθεί πάρα πολύ τα ποτάμια. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ από τα όσα επιτάσσει η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω αυτό το ερώτημα. Μιλήσατε για τα νητρικά άλατα. Έχουμε μερικά κράτη-μέλη τα οποία έχουν διαπιστώσει μια αύξηση της συγκέντρωσης των ε, νητικών αλάτων. Μπορείτε να μα δώσετε μια εικόνα για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Έχουμε, όπως είπατε, και ένα εφαρμογή. Τι συγκεκριμένο κάνετε με τις, ε, τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα και αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερα και οι συνάδελφοι. Αν χρησιμοποιείται και τις ε, νομικές διαδικασίες. Έχει αναφερθεί επίσης στη Γεωργία η διαδικασία του greening. Θεωρείτε ότι αυτό θα έχει κάποια επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων ή δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ελήψη άλλων ερωτήσεων δίνω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις. Και ιδιαίτερα στην κυρία Κεν. Ναι, γνωρίζουμε ότι η Δανία συζητάει. Ξανακοιτάζει τα μέτρα, τα αναθωρεί, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να δούμε ότι επιτυχάνονται οι στόχοι μέσω προγραμμάτων, μέσω μέτρων, σχεδίων που έχουμε στην Επιτροπή, που παίρνουμε στην Επιτροπή, μπορούμε να πούμε αν φτάνουν ή δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Τώρα βλέπετε βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο κύκλους. Στον πρώτο ήδη σχολιάσαμε και συζητήσαμε εκτενώς με τις χώρες μέλη και με τη Δανία. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι απόψεις μας. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο στάδιο και θα κρίνουμε από αυτό το κατά πόσο όντως ε, έχει φέρει σε πέρα στους στόχους της οδηγίας η Δανία ή όχι. Μόνο τότε δηλαδή θα μπορούμε να μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο και για το τι μέτρα ενδεχομένως θα πρέπει επιπλέον να ληφθούν. Με το λεκτικό συνέδριο και την έκθεσή του, την οποία βέβαια και διαβάσαμε πολύ προσεκτικά και τη συζητήσαμε μαζί τους, προσπαθούμε μαζί να βρούμε τρόπους θετικής ανταπόκρισης και να λάβουμε υπόψη μας πολλές από τις συστάσεις τους. Όχι για όλα τα θέματα, δεν θα μπορούσα τώρα να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες, πάντως είμαι σίγουρη ότι σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζουμε το ελεγκτικό συνέδριο στις συστάσεις του. Πάντως δεν είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντα, είναι στα χέρια των χωρών μελών. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες που πρέπει να πάρουν τα μέτρα, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι κρίνουμε κατά πόσο τα παίρνουν ή όχι. Και μετά μπορούμε να τους μιλήσουμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να τις πείσουμε τις χώρες μέλη, να τις βοηθήσουμε ώστε να λαμβάνονται τα σωστά μέτρα και σε περίπτωση ανάγκης τότε τους πάμε και στο δικαστήριο με την ε, διαδικασία επιπαραβάση Σας είπα ότι έχει ήδη συμβεί αυτό. Αυτά είναι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. είναι περισσότερο ένα θέμα που πρέπει να θέσετε στις χώρες μέλη. οι περιφέρειες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι με αυτά τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν ο καθένας όπως επιθυμεί. Αυτά. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Έχει να... του κύριου Βιτέμα. Θα δώσω και στην Επιτροπή βέβαια το λόγο για να απαντήσει και στην κυρία Μούλε. Ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε μιλήσει πολύ μέχρι τώρα για την οδηγία για τα νητρικά. Στα σχέδια διαχείρισης λεκανών, ο δεύτερος κύκλος προβλέπει ότι οι χώρες μέλη πρέπει να αξιολογήσουν που βρίσκονται όσον αφορά την κατάσταση και όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους βάσει οδηγίες για τα ύδατα. Πρέπει να εκτιμήσουν τον έλεγχο που κάνουν και να γίνονται οι έλεγχοι που χρειάζεται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται τα μέτρα. Όπως έχω πει και άλλη φορά στις απαντήσεις μου, πιστεύουμε ότι η οδηγία για τα νητρικά, εκείνη για τους οικότοπους, αποτελούν βασικά στοιχεία τις οδηγίες για τα ύδατα και χώρες μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτά τηρούνται. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι καταλαβαίνουν κατά πόσο φτάνουν ή όχι. Και τότε πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα. Είναι και αυτό απέτηση της οδηγίας για τα ύδατα. Έχουμε λοιπόν ήδη συζητήσει πολλά από τα μέτρα για να δούμε κατά πόσο λαμβάνονται στη Γεωργία ή αν είναι μέτρα τα οποία απορρέουν από τις απαιτήσει άλλων οδηγιών για τα πόβλητα για παράδειγμα και από εκεί και πέρα είναι στα χέρια των χωρών μελών και εφόσον καλύπτουν τα κενά και όντως καταλήγουν σε μια ικανοποιητική κατάσταση υδάτων, εμείς θα το διαπιστώσουμε αυτό και θα αντιδράσουμε βέβαια θετικά στα επόμενα σχέδιά τους διαχείρισης λεκανών. Για τη χρηματοδότηση έχω να κάνω μια παρατήρηση. Πρόκειται για την ανάπτυξη της υπαίθρου από τα εθνικά προγράμματα. Δεν πρέπει οι χώρες μέλη να ξεχνούν ότι διαθέτουν καλούς μηχανισμούς προκειμένου να βοηθηθούν να συμμορφωθούν με την οδηγία για την ποιότητα των υδάτων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρίουλα. Ούλα. Δεν θέλει το λόγο. Άλλος κανείς. Υπάρχει κανείς που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα που θέλει να ρωτήσει κάτι την Επιτροπή. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώς. Περνάμε στην επόμενη λοιπόν ερώτηση ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ήπεθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λέει η κυρία Διευθύντρια. Σας είπα από την αρχή ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τι ευρωπαϊκέ πρακτικέ και στι περισσότερε ε, περιπτώσει είναι αρνητικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα αλλά και την ακυρότητα του οικοσυστήματο. Διότι έχουμε αρκετά στοιχεία ε, όσον αφορά τι εκθέσει ε, τι εφαρμοστικέ Καθώ επίση και στι εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλον που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Προφανώ και αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα επίση προκαλούν κάποιε δαπάνε. Τις δαπάνε αυτές τις φέρουν οι κύριοι των γεών αυτών η γεωργία αλλά βέβαια και όλη η κοινωνία γιατί όταν μιλούμε για ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να μπορεί να το πιει ο κόσμος επίσης έτσι υπάρχει ευξημένος κίνδυνος πλημμύρα και έχουμε μείωση αυτών των κινδύνων ε, με διάφορα μέτρα που βοηθούν να ε, ανασχεθεί αυτή η διάβρωση του εδάφους και επίσης έτσι ε, λέμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, για τη γεωργία ε, και για την ε, κοινωνία γενικότερα. Τώρα, τι θα κάνουμε για αυτό. Ο κόσμος της γεωργίας, ο χορτικός κόσμος, σαφώς και ζητεί το να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Και, πολύ συχνά, αυτό ε, επίσης μας ε, οδηγεί ε, στο να λάβουμε υπόψη το αριθμό και το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μην ξεχνάμε ότι η γεωργία παίρνει το 40% του προϋπολογισμού, οπότε θα πρέπει και οι γεωργοί να προσαρμοστούν στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Γιατί ακριβώς αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Τα χρήματα υπάρχουν για τους δύο πυλώνες της ε, αγροτικής γεωργικής πολιτικής. Οπότε και οι γεωργίες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν το ότι κάνουν αυτό που πρέπει. Όμως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει κάποια πιο συντονισμένη προσπάθεια ε, όσον αφορά τις πληρωμές της γεωργικής πολιτικής, όσον αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα και οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο οι γεωργοί δικαιούνται κάποιων αμέσων πληρωμών εάν έχουν λάβει τα συγκεκριμένα κατάλληλα μέτρα. Αν έχουν δηλαδή ε, κάποιο είδου ε, φράγματα, κάποιες ζώνες ανάσχεσης των υδάτων, ε, έχουν ενεργήσει έτσι που να είναι ασφαλή, ασφαλές το επιβάλλον, αν έχουν κάποιους ε, φράκτες από θάμνους, ε, οπότε και όλα αυτά ε, την χάνουν υποστήριξης από τις οικονομικές ενισχύσεις. Επομένως δεν κάνει μοναχικό αγώνα ο καθένας. Υπάρχουν πόροι και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Και ακριβώς στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου γιατί και τα κράτη-μέλη πρέπει να επεξεργαστούν τα δικά τους προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Και εμείς τα λαμβάνουμε αυτά τα προγράμματα, τις προτάσεις στη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία. Διαπιστώνεται επομένως ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές ε, είναι ανίδεα του τι προβλέπεται. Γιατί υπάρχουν αυτά τα μέτρα, ε, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν τη χρηματοδότηση ε, και όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε, τις οδηγίες για τα αζωτούχα λοιπάσματα, για, για την οδηγία πλαίσιο, για οτιδήποτε. Οπότε και εμείς ε, εντατικά συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους της Γεωργίας. Και έτσι τα κρατημέλη θα πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα ότι λεφτά υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται προσπάθεια να τους τα πούμε πολλές φορές και ε, αναρωτιόμαστε μα γιατί δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν ξέρουν ότι τα χρήματα αυτά διατίθενται. Γιατί υπάρχουν οι πόροι, προβλέπονται, αλλά δεν απορροφώνται. Επομένως θα πρέπει να γίνει περισσότερη ενημέρωση και θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν. Επίσης, έχουμε κάποια έγγραφα όπου παρέχονται κάποιες κατευθυντήριες για κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δυσανάλογα όσον αφορά το όφελο σε σχέση με το κόστος. Θα μπορούσαν αυτά να ε, χρησιμοποιηθούν όπως ας πούμε κάποιο είδους ε, βιωσιμότητα τεχνολογική σε σχέση με το κόστος, όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και έτσι να εξασφαλιστεί ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο δεν θα χρησιμοποιηθεί Έχουμε επίσης τις διατάξεις της οδηγίας για τα ύδατα που και αυτά συντρέχουν κάποιες φορές αλλά χρειάζεται κάποια διαδικασία διαφάνειας ότι θα πρέπει δηλαδή όλα να δικαιολογούνται, θα πρέπει να τεκμηριώνονται και εμείς επίσης θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη απορροφούν καλύτερα αυτά, αυτές τις ενισχύσεις που προβλέπονται ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει οικονομική υποστήριξη των ε, γεωργών και ότι θα συμμορφώνονται με τους στόχους της οδηγίας για τα ύδατα και ταυτόχρονος θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές θα διαχειρίζονται τα προγράμματα ξέροντας ότι υπάρχουν λύσεις και μέτρα και επομένως οι αρχές αυτές θα πρέπει να ενημερώνουν ε, τους εμπλεκόμενους στη χώρα τους. Και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Μήπως υπάρχουν ερωτήματα από τους συναδέλφους. Όχι δεν υπάρχουν. Τότε μπορούμε να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Από την κυρία Ριβάζη για τα φάρμακα στα νερά ή τα νερά στα φάρμακα και δεν απαντήσει και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολύ καιρό ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Έχουμε μια μελέτη που ε, ζητήσαμε να εκπονηθεί και παρουσιάστηκε πέρσι τον Ιούνιο, συζητήσει σε ένα εργαστήριο τον Σεπτέμβριο, συζητήσει το 2014 όπου οι σύμβουλοι μας είχαν δώσει κάποιες εναλλακτικές λύσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε τα φαρμακευτικά στα νερά. Και στρατηγικές ή τουλάχιστον ενάψματα για στρατηγικές που θα μπορούσε η Κομισιόν να αντιμετωπίσει για να καλύψει τη, τα πετούμενα από την οδηγία για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας για το θέμα αυτό για να δούμε τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε. και ας συνεχίσουμε να προχωρούμε με τον δρόμο με τον οποίο συνεχίζουμε τις συζητήσεις αυτές προς την κατεύθυνση της περαιτέρω συνέχισης των συζητήσεων εσωτερικά με τις υπηρεσίες μας και με τους διάφορους εμπλεκομένους. Θα πρέπει να δούμε πότε τελικά θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε μια τέτοια στρατηγική και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εντοπίζει τα μέτρα που απαιτούνται σε επίπεδο δυνητικό. Εάν προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, τότε η στρατηγική θα πρέπει να προβλέπει αυτά τα μέτρα και κάθε πολιτική, όπως ξέρετε, υπόκειται σε εκτεταμένη έκθεση αντικτύπου. Θα χρειαζόμαστε λοιπόν χρόνο για να μπορέσουμε να έχουμε μια διαβούλευση σε σχέση με τα θέματα αυτά. Εν τω μεταξύ, ο νέος κατάλογος για τα θέματα που πρέπει να οδηγήσουν σε εποπτεία από την Κομισιόν θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες και αυτό θα περιλαμβάνει και την παρακολούθηση των φαρμακευτικών ουσιών που βρίσκονται στον κατάλογο και προέρχονται από τη διαπραγματεύση για τα πρότυπα ποιότητα του περιβάλλοντος. Τα αντιβιωτικά λοιπόν αυτά συγκεκριμένα. Η επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος ξεκινάει τώρα και αφορά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τον δυνητικό κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκύψει από, άλλε, από φαρμακευτικές ουσίες και άλλους μικρορύπαντες πολύ σοβαρά και είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στη συνέχιση του έργου μας και όταν, όταν τελειώσουμε θα σας τα διαβιβάσουμε όλα με απόλυτη διαφάνεια σε όλους τους άλλους εμπλεκομένους. Κυρία Ριβαζή, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά δεν με ικανοποιεί και ιδιαίτερα. Γιατί βάσει της οδηγίας του 2013 η Κομισιόν έπρεπε να έχει εκπονήσει μια στρατηγική προσέγγιση για τη ρήπανση των υδάτων μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του 2015. Κάνετε νέα πράγματα όπως για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Σας ζητάει το Κοινοβούλιο να εκπονήσετε μια στρατηγική. Θυμόσαστε, το 2013 είχαμε κάνει αυτό για τους ε, διαταράκτες. Έπρεπε να την έχετε αυτή τη στρατηγική το 2015 και λέτε ναι, μα θα κοιτάξουμε αν υπάρχουν προβλήματα κτλ. Μα, κοιτάξτε. Έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα κατάλογο των ουσιών που προέρχονται από φαρμακευτικά σκευάσματα και που ξέρετε ή που μπορείτε να διαπιστώσετε ότι θα οδηγήσουν σε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Αν έχετε αυτό τον κατάλογο, εμεί μπορούμε να πιέσουμε τα κρατημέλη μελη να σεβαστούν αυτόν τον κατάλογο. Αν όμω αφήσετε τα κρατημέλη να κάνουν αυτό το έργο, θα πούν τα κρατημέλη μα δεν έχουμε επιστημονική εμπειρογνώμηση, δεν κάνουμε τίποτα. Σα έχει δώσει λοιπόν μια γραμμή το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο και δεν την ακολουθείτε η ιστορία της Volkswagen. Αν βλέπετε, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τοξικότητος είναι πεπαλαιωμένα. Κάνουμε κάτι και για, και για τα βακτηρίδια και εκεί πρέπει να δούμε ποια είναι η τοξικότητα που επιφέρουν τα βακτηρίδια στο πόσιμο ύδωρ. Είναι καιρός να επανεξετάσετε αυτά τα, αυτές τις δοκιμασίες. Για την Volkswagen, ναι, τα τεστ δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και με το πόσιμο είδα. Πρέπει να προτείνει η Κομισιόν νέα τεστ για τι χημικέ ουσίε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η προβληματική των ενδοκρινικών διαταρακτών που βρίσκει κανεί στο είδωρ και έχουμε και τα κοκτέιλ που κάνουν μεταξύ τους οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και δεν κάνετε τίποτα για αυτά. Έχουμε βρει πάνω από 160 ουσίες που προέρχονται από φάρμακα στα ύδατά μας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Λέτε ότι είναι πιο οικολογικό να πίνει κανείς το νερό της φρύσης παρά να αγοράζει νερά από την αγορά και εκεί πέρα κολυμπούν και κάνουν πάρτι όλες αυτές οι ουσίες. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να δράσει πιο μεγάλη προδραστικότητα, να κάνει προτάσεις όταν έχετε μια καταληκτική προθεσμία, σεβαστείτε την, ε, αν μπορώ να σας το πω, ούτως. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Και πάλι η Κομισιόν για να αντιδράσει. Ναι, ναι, σας άκουσα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι αποστερημένο πολυπλοκοτήτων σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία βρίσκονται στο είδωρ. Έχουμε μιλήσει με τις αρχές των υδάτων και ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα αυτού του είδους ένα πρόβλημα όμως το οποίο ξέρω ότι δεν οδηγεί σε προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία είναι αυτό γιατί βρίσκονται σε μια ποσότητα η οποία είναι κάτω από τα θεσπιστέντα όρια από τις νομοθεσίες μας σε ό,τι αφορά το πόσιμο ειδό και δεύτερον προς το παρόν εμείς παρακολουθούμε τις ε, τάσεις που αναδύονται γιατί μπορεί να αυξάνονται οι ουσίες αυτές προσπαθούμε να δούμε αν εξαλείφονται ή όχι. Υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να τις εξαλείψουν, αλλά αυτό επέχει και ένα συγκεκριμένο κόστος. Θα πρέπει να πληρώνουν και οι καταναλωτές για την εξάλληψη αυτών των αγαθών βακτηριδίων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ρίζα του, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, με τους άλλους εμπλεκομένους. Ξέρουμε ότι μια σειρά από κράτη-μέλη ακολουθούν ενεργά μια στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Είμαστε σε επαφή μαζί τους, συζητάμε, αλλά προς το παρόν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και είμαστε καθυστερημένοι, αλλά είμαστε καθυστερημένοι επειδή είναι πολύ πλοκό το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πάμε στην τελευταία ερώτηση για σήμερα. Αριθμός 8. Κύριο Πεντιτσίνη, η FDD. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. The honorable member when he mentioned it uh, previously. Α, ναι, ναι. Προηγουμένως τα είπε ε, ο κύριος βουλευτής και εμείς. Απαντήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την γραβή ερώτηση που είχε υποβληθεί και εκείνη για το ίδιο θέμα, διότι πρόκειται για τα πλαίσια της συνεχούς ερεύνης και αυτό το τονίσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αξιολογήσει όλα τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει οι Ιταλικές Αρχές και έτσι ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον συνάδουν τα μέτρα αυτά της ε, ε, λίμνης Πέτρου Ζήλου με τα όσα προβλέπει η οδηγία. Και επομένως δεν είναι το θέμα του ότι αγνοούμε του τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θέμα και πρέπει να ρυθμιστεί και αντιμετωπιστεί. Σας είπα τι κάναμε ακριβώς, αυτό κάναμε, αλλά επίσης ήδη βρισκόμαστε στην διαδικασία αυτής της έρευνας για την οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε όσο αυτή εξελίσσεται. Πάντως σας επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για μια πιλωτική υπόθεση. Προχωράμε. Έχουμε επαφές με τις τελικές αρχές και επίσης έχουμε τώρα ε, και κάποιες επιπλέον πληροφορίες τις λάβαμε τον Απρίλιο και αξιολογούμε αυτές τις πληροφορίες και επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης πρόκειται να αναλάβουμε δράση αναλόγως. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά νομίζω ότι ο κ. Πιτετζίνη θέλει να σας πει κάτι. Ναι, ναι, ναι, μια, μια απάντηση σύντομη. Έχουμε πληροφορίες που οι τοπικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την περιοχή έχουν δώσει ότι δηλαδή έχουν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποιες ε, τιμές αυτών των βαρέων μετάλλων και των αθράγων που είναι πολύ παραπάνω από τις ουρακές τιμές που προβλέπονται κατά ε, πολλές, πολλά δεκαδικά ψηφία τέλο πάντων και οι πολλές δεκάδες. Οπότε τι θα γίνει τελικά. Ε, έγινε η διαδικασία επιπαρέμβαση και δεν απέδωσε τίποτα. Μα τελικά όμως το, την ύφη την πληρώνουν οι πολίτες και παθαίνει η υγεία τους. Δηλαδή είδαμε ότι η μέθοδος που ακολουθήσατε δεν αποδίδει. Και εμείς πρεσβεύουμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να συζητηθούν κάποια νέα, περαιτέρω μέσα για να παρέμβει κανείς εκεί σε αυτό το, χώρο. Η διαδικασία ενώπιν του δικαστηρίου δεν αποδίδει. Όταν υπάρχει κάποια διοικητική αρχή η οποία ε, επιβάλλεται από τα μεγάλα λόμπι που τους υποστηρίζουν τις ε, προεκλογές εκστρατείες ή και κάποια βιομηχανικά συμφέροντα. Οπότε μετά τους χωστάνε χάρη και οι αρχές αυτές ε, ανταποδίδουν τη, τη χάρη αυτή. Που, οπότε και γίνεται αυτή όλη η μόλυνση. Και όταν γίνεται επομένω αυτή η αγωγή η παραβάση δεν κάνει τίποτα. Όποιος μολύνει πληρώνει. Δεν ισχύει αυτή η αρχή κατά αυτόν τον τρόπο και πληρώνουν δύο φορές οι πολίτες. Να ποιο είναι το αληθές πρόβλημα. Γι' αυτό εμεί λέμε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Γιατί το να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία η παραβάση δεν ωφελεί, γιατί είπαμε ότι δεν ωφελεί. Και πληρώνουν και τα έξοδα οι πολίτε. Σα ευχαριστώ. Πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Εκπλήσουμε κάπως. Όχι, όχι, όχι, είναι ε, ε, διαδικασία πιλωτική υπόθεση. Δεν είμαστε στη διαδικασία αγωγή ή παραβάση. Και κάθε φορά που ξεκινά μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να ισχύσει ο κανόνα τη υπεράσπιση. Δηλαδή θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε κάτι στο κρατό μέλο των εμπλεκόμενων και αυτό θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στι εμπλεκόμενε αρχέ οι οποίε έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν ε, εαυτού, δηλαδή να πούνε ότι υπάρχει αυτό και κάναμε αυτό και λοιπά και λοιπά. Οπότε και τελικά ε, εάν όλα αυτά είναι βάσιμα πάμε στο δικαστήριο. Είναι αυτή η διαδικασία η οποία έχει αποδώσει. Είναι ε, μακρά διαδικασία αλλά ε, χρειάζεται να γίνει, δικαιολογείται. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις μιλούμε και συνομιλούμε απευθείας με τις εθνικές αρχές, με τους ομολόγους μας. Ακριβώς όπως τα πλαίσια της οδηγίας για τα ύδατα. Βοηθούμε τις εθνικές αρχές. Και όσον την ερμηνεία ορισμένων άρθρων της ε, οδηγίας. Ε, όταν μιλούμε τώρα για κάποιες οριακέ τιμές, τι να πούμε, τι να ερμηνεύσουμε. Τους λέμε συμμορφωθείτε με αυτές τις οριακές τιμές για τον αέρα, για τα νερά κλπ. Και, και φτάνω σε αυτό που θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία μας περιγράφεται είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Το κρατός μέλος θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και έτσι να εξασφαλίσει ότι ο κόσμος αυτοί που ζουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος είναι ασφαλής από ρυπάνσεις, μολύνσεις που ενδεχομένως υπάρξουν. Δεν μπορούμε άμεσα να κάνουμε τίποτα. Μόνο σε πολύ πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν έχουμε μέσο παρέμβασης. Και ευτυχώς που δεν μπορούμε να παρέμβουμε γιατί αυτό θα ανέτρεπε όλη την ισορροπία το, το, το, τον αρμοδιο, του πλέγματος αρμοδιοτήτων κομισιών, κράτους μέλους κλπ. Η εφαρμογή των κειμένων νόμων είναι πάντα εθνική αρμοδιότητα. Οπότε, πραγματικά, τι να σας πω. Τι να σας πω, μόνο να, να απευθυνθώ σε εθνικές αρχές και να τους πω να κάνουν αυτό το οποίο θεωρούν ότι είναι αναγκαίο, ούτως ώστε το περιβάλλον και ο κοσμάκης είναι ασφαλής. You uh, με, Πρόεδρε. Κάτι μου ε, πρότεινε τώρα ο, ο συνάδελφος. Και σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να ενεργήσετε από πλευράς ε, δικονομίας. Γιατί εκεί ξεκινά η διαδικασία αυτή στις περισσότερες, σε πολλές τέτοιες υποθέσεις. Πρώτα, σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υποβάλλονται καταγγελίες, όποτε και εκεί προβλέπεται η δυνατότητα η Εθνική Ένωμη να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή της οδηγίας γίνεται Μόνο όταν αυτό δεν αποδώσει τότε κανείς προσφεύγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πιένσω στη διαδικασία. Thank you very much. I think... Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε εδώ να κλείσουμε αυτό το τμήμα της συνάντησή μας. Οι άλλες ερωτήσεις θα πάνε για την επόμενη τέτοια συνάντησή μας. Ζητώ από τους Προέδρους, τον κύριο Σικέσκι, Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης να έρθουν εδώ μαζί μου στο Προεδρείο. Και τα μέλη των Επιτροπών αυτών ας έρθουν και ας καθίσουν προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ας διακόψουμε δύο λεπτά. Δύο λεπτά διακοπή.